Dear colleague, we open the seat. Thank you to be here and to... Καλημέρα συνάδελφοι, καθίστε, ευχαριστώ που ήρθατε. Καθίστε ξαναλέει η Πρόεδρος. Να συνεχίσω στα Ιταλικά. Ωραία. Καλώς ορίσατε. Σήμερα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Περιμένω λίγο να Εντάξει. Έλεγα ότι έχουμε μια μέρα πολύ φορτωμένη και το πρωί το απόγευμα και όλοι οι συναδελφοί θα πρέπει να έρθετε και το απόγευμα. Γιατί το απόγευμα έχουμε μια κρόση πολύ σημαντική. Οπότε και εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες. Επίσης, για να δούμε τώρα το πρώτο μας θέμα, η έγκριση της ημερήσιας ε, διάταξης, υπάρχει ένσταση, προχωράμε, δεύτερο τμήμα, τα πρακτικά της 14, 15, 21 Σεπτεμβρίου, ούτε εδώ ε, έχουμε ένσταση, οπότε πάμε στο επόμενο σημείο και όσον αφορά τη διερμηνία, σήμερα Έχουμε προσβία από γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά, φιλανδικά, τσεχικά, εστονικά, σλοβακικά, σλοβενικά, μαλτέζικα, πορτογαλικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και επίσης για την ακρόαση έχουμε σουηδικά αλλά και ολλανδικά. Οι συνεδρίες μεταδίδεται στο ίντερνετ και η πρώτη ανακοίνωση που έχω είναι το εξή. Έχουμε τα Lux Prize και είπαμε ότι αυξάνεται η σημασία τους, υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία, συγγνώμη, συμμετοχή από όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να θυμάστε ότι πρόκειται για το μοναδικό, μοναδικό βραβείο όπου οι ίδιοι είμαστε η κριτική επιτροπή και οι συνάδελφοι συμμετέσχουν και διάλεξαν τους τρεις φιναλίστ. Του χρόνου θα είναι η δέκατη επέτειος, οπότε θα γίνει η ορταστική πανηγυρική ε, διαδικασία. Οπότε και η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο ε, πρόκειται έτσι να συμβάλλει στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο και στη δουλειά των νέων πάνω σε αυτά. Επίσης έχουμε τις εκδηλώσεις του Καρλό Βιβάρη και εκεί θα έχουμε πολύ σημαντικές ε, εκδηλώσεις από πλευράς καλλιτεχνικής και γενικότερα πολιτιστικής για όλη την Ευρώπη θα ζητηθούν θέματα και της κρίσης, ο ε, αντισημιτισμός, ολοκαύτωμα, όπως επίσης και κάποια άλλα θέματα γραφειοκρατίας. Έχουμε το θέμα του πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, ε, θέματα για τους Ρώμ, ε, την μετάβαση από την παράδοση στον νεοτερισμό, στον φροταδιόν των γυναικών και έχουμε κάποιες Ταινίε των φιναλίστ. που μερικά εξ αυτών έχουν παρουσιαστεί και για Όσκαρ. Ράμς, το πρώτο Ισλανδικό έργο που κατέβηκε στο Λουξ, το Χάι Σαν, μια συμπαραγωγή από την πρώην Ιουγκοσλαβία, από Ουγγαρία, στο Σάουλο, είναι για το Auschwitz, συγκλονιστικό και αυτό κατέβηκε για Όσκαρ. Και Έχουμε και το Mustang ε, γαλλικό, και στην Τουρκία από μια νέα τουρκάλα σκηνοθέτη. Αυτά κατέβηκαν και ε, στην, στο φεστιβάλ της Βενετίας, οπότε και θα πρέπει βέβαια να πούμε μπράβο σε αυτά τα φεστιβάλ τα οποία προβάλλουν ε, τα έργα που συμμετέχουν στο Λουξ. Και ευχαριστούμε τους συναδέλφους λοιπόν οι οποίοι με μένα ε, συμμετέσχουν στις εκδηλώσεις εκείνες. για την προβολή αυτών των έργων και στη Βενετία και έχουμε επομένως τους επομένως 28 πρέσβεις του Λουξ είναι αυτοί οι νέοι σκηνοθέτες προέρχονται ο καθένας από άλλο κράτος μέλος και συμμετέχουν δυναμικά και σε αυτό το σεμινάριο το οποίο γίνεται. Και αυτοί φέρνουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη διάδοση του Λουξ. Έχουμε επομένω του τρει φιναλίστ, οι οποίοι με ψηφοδική σα θα κρυθούν. Το Μάσταγκ, όπω είπαμε, την Τένι Γκάμ. μια τουρκάλα σκηνοθέτηδα, ε, το ροκ επίσης συγκλονιστικό το έχω δει ε, μιας βουλγάρας σκηνοθέτηδας Κριστίνα Γκρόσεβα και του Πάτερ Βαλκάνοφ είναι ελληνοβουλγαρική και το Μετεράνια του Σκαρπινιάνο μια συμπαραγωγή ευρωπαϊκή με τη συμφωλή του Sundance Film Festival των ΙΠΑ. Είναι τρεις ταινίες ε, ψηλής ποιότητας και ευαισθησίας. Στις 19 Οκτωβρίου θα αρχίσει η κρίση και μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχετε κρίνει. Από τις 19 Οκτωβρίου είτε με βίντεο in demand είτε με άλλους τρόπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους υπαλλήλου που έχουν ασχοληθεί με αυτό. Είναι οι υπάλληλοι του Γραφείου της Επικοινωνίας του Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επομένω όλα αυτά τα έργα ε, θα διατίθενται και όποιος θέλει μπορεί να τα παρακολουθήσει. Οπότε μπορείτε και όχι μόνο να ψηφίσετε αλλά μπορείτε και να τα διαδώσετε στα, στις χώρες σας ε, αυτά τα έργα και έτσι να ανακατευτούν περισσότεροι από τον κόσμο να μάθει εκείνη η γνώμη δηλαδή. Και βλέπουμε, λέμε διάφορα, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά υλοποιούνται σε αυτού του είδους την, την αντιπροσώπευσή μας σε αυτόν τον διαγωνισμό με αυτά τα έργα. Και έτσι θα μπορέσουμε αυτά τα έργα να τα προβάλλουμε σε όλη την Ευρώπη και αυτό μπορεί να γίνει από τις αντιπροσωπείες, τα γραφεία τέλο πάντων του Κοινοβουλίου σε όλη την Ευρώπη. Και θα γίνει η πανηγυρική τελική ε, τελετή στις 25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Παρουσία του Πρόεδρου Σούλς και των τριών φιναλίστ που θα είναι εκεί. Και εκεί θα ανακηρυχθεί ο νικητής του διαγωνισμού. luxprize.eu κάθετος vote. Είναι το site στο internet μπορείτε να ψηφίσετε. Και επίσης μπορείτε να δείτε αυτά τα έργα στον χώρο Γιβούντι Μενοχήν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Στις 11 Νοεμβρίου δε θα γίνει μια προβολή του Μεντιτεράνια στις 7.30 το απόγευμα. Και αυτό θα γίνει ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Και κατόπιν στις Βρυξέλλες, στο Μποζάρ, θα έχουμε τον Σκαρπινιάνο, τον σκηνοθέτη. Θα συμμετέχει το Σεφεστέλ της Μπρατισλάβας, της Βίλης, το Φόρουμ Ημάρ του Βαρισιού, το Cinema City της Λισαβόνας και στο πειραματικό φεστιβάλ της, ε, του Βουκουρεστίου. Και οπότε και αυτό θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θα αφορά την προβολή στην Ευρώπη αυτού του διαγωνισμού. Οπότε έτσι σας θυμίζω ότι και το ΑΡΤΕ πρόκειται να προβάλλει την εκδήλωση. Η γραμματεία του Λουξ οι φίλοι Ρωσοί. Ποιοι είναι. Εδώ είναι. Α, ήταν εδώ πριν από λίγο. Και άλλοι συνάδελφοι πρόκειται ε, να έχουν όλο το υλικό που χρειάζεται. Και ευχαριστώ και τον Μπόγκταν Βέντα, τον συνάδελφο, γιατί και αυτός παρακολούθησε όλες αυτές τις συζητήσεις που έγιναν και στα προηγούμενα φεστιβάλ και για τις προβολές των έργων Οπότε είναι σημαντικό του χρόνου που θα γίνει αυτή η επέτειος να συζητήσουμε συντολιστές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε τη σημασία του βραβείου. Οπότε, παρακαλώ, δείτε τα έργα και ψηφίστε. Γιατί έτσι αποδεικνύονται οι για τον πολιτισμό με το να συμμετάσχουμε εμείς οι να ψηφίσουμε περισσότερο και από πέρσι. Και έτσι το μήνυμα θα είναι πιο αποφασιστικό το φετινό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ε, ερωτήσεις, αλλιώς πάμε στο τέταρτο σημείο που έχουμε που είναι ψηφοφορία. Έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε μια σημαντική έκθεση. Προέρχεται από τον συνάδελφο Κρασνοντέμψικη. Τον ευχαριστούμε και αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο αν θέλει. Έχουμε 98 τροπολογίες. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τη συνεργασία που είχαμε. Ήταν πραγματικά πολύ αρμονική και αγαστή και ελπίζω ότι θα υπερψηφίζουμε την έκθεση. Δεν είχαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ μας και διαφωνίες. Κάποιες μικρολεπτομέρειες αφορούσαν περισσότερο. Και νομίζω ότι μια και ήταν κοινό ο στόχο, απλώς προσπαθούσαμε να βρούμε τις κατάλληλες διατυπώσεις για να τον αποτυπώσουμε με τρόπο που θα ικανοποιεί όλους του συναδέλφους. Περιμένω την ψηφοφορία. Ωραία. Ε, οπότε, επί τη βάση όλων αυτών, πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά στην ψηφοφορία. Για πέστε μου, έχετε όλη την κάρτα, για να δω κι εγώ. Scusate un momento, succede. Sorry, but I'm afraid of to have to left my... Συγγνώμη, ε, εγώ ξέχασα στην ε, Ολομέλεια τη δική μου κάρτα. You? No, no, the card. Δεν κατάλογο ψηφοφορία. Την Χειρότερο, την κάρτα μου έχω ξεχάσει την Ολομέλεια. <laughs> the card. It normally that uh, uh, doesn't happen, but sometimes. Ε, καμιά φορά συμβαίνει, σπανίως όμως. Αν δεν σας πειράζει να ψηφίσω υπογράφοντας, έτσι κι δεν είναι μυστική ψηφοφορία, με ανάταση της χειρός δηλαδή. Ωραία. Ουνο. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, παραθμόν ένα του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Όχι, α, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο 9. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Α, αποχές. Να το ξανακάνω. Υπέρ. Για το 9, για το 9. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτω. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. πέρας. Approved. Approvato. Emendamento 12. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά Ας κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Χες εγκρίνεται 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Και το 37 κάνουμε παλίτες. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν δεν σηκώσταν και το λοιπόν ψηφίζουμε τώρα για το 39. Επαλήθευση για το 39. Υπέρ, ε, έναρξη τέλος της εφορίας. Α, ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Απορρίπτεται. Ε, κάποιοι σηκώσαν εργατά χέρια, τέλο πάντων. 40 για την παράγραφο 3 α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 του εισήγητη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στο συμβαστικό 7 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στο 64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 απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 του εισηγητή είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά ξανά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο Ψηφίζουμε. Πέρας. Με δύο ψήφους διαφορά εγκρίνεται. Όχι. Δεν το βλέπετε. 14, 12. Και δύο αποχές. 83 υπέρ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 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 το εισηγητό και πάλι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνει. Παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία. Everybody's vote? Okay. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 22 ψήφισαν υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κρασνοντέμσκι. Thank you also to Shadow Rapporteur, to ε, Ευχαριστώ και τους και ηγητές και, όσους, και όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή. Και τώρα πάμε παρακάτω για κάτι το υπέροχο. Γιατί έχουμε τώρα σε επαφή με κάποιους νέους που οικοδομούν την Ευρώπη και αυτή τη φορά επομένω τα μαντάτα δεν είναι κακά. Γνωρίζετε ότι έχουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων με κάποιους ε, εξέχοντες συνομιλητές είναι οι οκτώ νέοι που προέρχονται από τις ε, εθνικές ομάδες που κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάνου που ξεκίνησε το 2009. Όχι, 2008. Είναι κοινή πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, του Διεθνούς Ιδρύματος Καρλομάνου Καλώς όρισαν οι νέοι βραβευθέντες, να οι πρώτοι τρεις. Λουξεμβούργοι. ονομάζεται Real Time W, 1 Δεύτερον, από τη Γαλλία, Fronteras, European Border, σαρφρέμ και το τρίτο από την Αυστρία. Είναι το ε, Social Soccer Cup και επίσης έχουμε και από την ε, Κύπρο ε, entrepreneurship, the solution και στην employment, επιχειρηματικό πνεύμα και info actualidad από την Ισπανία. Από Χόρχε Καναβέρας και Κριστίνα Αλόνσο Γκαρσία. Καλώς ορίσατε. Κοιτάξτε, να κάνουμε μια κοινωνική φωτογραφία γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η στιγμή και για εσάς και για εμάς. ελπίζουμε ότι πρόκειται για μια περιπέτεια υπέροχη το να συμμετέχετε εδώ ε, και επίσης το ότι έχετε κερδίσει και ότι μπήκατε στους φιναλίστε οπότε και εμείς εδώ με χαρά μας σας υποδεχόμαστε και τώρα με τη σειρά για τα λεπτά να πάρετε το λόγο να μας παρουσιάσετε το, το δημιουργήσατε και κατόπιν να κάνουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ είμαστε περίεργοι να μάθουμε τι έγινε, πώς τα φτιάξατε αυτά Οπότε, πρώτα-πρώτα, πάμε από το τρίτο στο πρώτο, άρα να πάρει πρώτο το λόγο η, η Γαλλία, κύριε Σαραφρέν. Dov'è? Eccola. Prego, a lei la parola. Ehm, bonjour, mesdames et messieurs les députés européens. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτέ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας, ε, τα project μας, μεγάλη τιμή για μας. Όπως ε, βλέπετε, το δικό μας project αφορά τα σύνορα. Διακόπτει η Πρόεδρος. Μπορούμε λίγο να χαμηλώσουμε το φωτισμό, παρακαλώ. Oui, alors c'est δεν ε, περιγράφει τα σύνορα το project μας, ε, αλλά ουσιαστικά παρουσιάζει μερικές προσωπικές ιστορίες ε, που τις βίωσαν οι άνθρωποι είτε με τα σύνορα είτε στα σύνορα. Πρόκειται για ανθρώπους που ταξιδεύουν και έχουν μια προσωπική εμπειρία, ένα προσωπικό βίωμα με τα σύνορα. Γι' αυτό και λέγεται Ευρωπαϊκή Μεθόριος, η Ευρωπαϊκή Συνοριογραμμή. Βλέπετε το site μας, το πιο σημαντικό τμήμα αφορά τα ρεπορτάζ που κάνουμε. Ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια το σχέδιό μας ε, στην Ευρώπη που βρεθήκαμε μερικοί φίλοι στην πλατεία του Λουξεμβούργου και σκεφτήκαμε γιατί δεν κάνουμε ένα site με ένα ρεπορτάζ που θα παρουσιάσει τα προσωπικά βιώματα των κατοίκων της Ευρώπης. Πάνε τρία χρόνια από τότε και δημιουργήσαμε ένα μικρό σύλλογο 40 ατόμων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας σε ρεπορτάζ στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και σε άλλες ακόμη γλώσσες, γιατί δεν έχουμε γλωσσικούς περιορισμούς. Τα βιώματα αυτά, οι ιστορίες αυτές είναι γνήσιες, ε, σημαντικές, μερικές φορές ε, θλιβερές, άλλες φορές διασκεδαστικές. Δεν ε, έχουμε εξακριβώσει την γνησιότητά τους, πάντως επιμένουμε στην αρχή της ανοχής και κάνουμε λογοκρισία σε ρατσιστικά, ξενοφοβικά ή άλλα σχόλια που δείχνουν μία έλλειψη ανοχής. Στις τρεις πρώτες γραμμές ε, βλέπετε τον Κλάρτ, τον Ζουλιαν Ποντρί και δικούς μου φίλους, τον κύριο Χάνεμαν. Έχουμε μερικούς ε, πιστούς ε, οπαδούς αυτού του σχεδίου. Πρόκειται για ανθρώπους που ε, είτε κατάγονται από την Ευρώπη είτε από άλλες χώρες, τρίτες. Όπως σας είπα είμαστε γύρω στους 40 στην ομάδα μας. Πάνω από 9 χώρες συμμετέχουν ε, στο ρεπορτάζ 17 ε, σύνορα και 4 χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλγερία, Μαρόκο, Αζερβαϊτζάν και μάλιστα μερικά ρεπορτάζ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, πραγματικά προσπαθούμε να κάνουμε αυτήν, αυτό το σύλλογό μας ένα φυτόριο διασυνοριακών βιωμάτων. Κάθε μήνα έχουμε ένα ρεπορτάζ και προβάλλουμε μια συγκεκριμένη προσωπική ιστορία, κάπως πιο πρωτότυπη, τουλάχιστον διαφορετική. Αυτή τη φορά έχουμε την Αντέλ που κάνει το ταξίδι Μασαλία-Αλγέρι και πάντα έχει προβλήματα στα σύνορα σταματάει σε ένα μπιστρό, αγοράζει τρόφιμα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική μερικές φορές. Αρκετά απολαυστική ιστορία της. Παρακαλώ σας παραπέμπω να την ε, να κοιτάξετε το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε εμείς πριν από τέσσερα χρόνια στις Βρυξέλλες όταν αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το project. Επίσης ε, έχουμε μία κατηγορία όπου άνθρωποι θέλουν με φωτογραφίες να μας παρουσιάσουν το ταξίδι. Δεν χρειάζεται να έχουν και κείμενο. Κάποιος που ταξιδεύει κάθε μήνα στη Μόσχα μας παρουσιάζει τους συνεπιβάτες του στο τρένο που κάνει τη διαδρομή Βερολίνο-Μόσχα, για παράδειγμα. Ένας Γερμανός. Επίσης έχουμε κάποια δύσκολα σύνορα, όπως το Αχτοκστράτ Γκρέντσε. Δείχνει ε, τέτοιες καταστάσεις πιο φιλικά σύνορα, πιο συμπαθητικά, Σλοβενία-Ιταλία. Ο Τζοβάνι μας παρουσιάζει αυτά τα σύνορα. Ή έχουμε πιο περιφερειακά σύνορα, είτε στη Γερμανία, είτε στην Ιταλία, το Τραστέβερε, όπου οι ε, κάτοικοι του Τραστέβερε, της τη αυτής της ε, Ρώμης, ε, ισχυρίζονται ότι εκεί βρίσκεται η καρδιά της Ιταλικής κουλτουρα Αυτά λοιπόν, έτσι κάνουμε τα ρεπορτάζ. Βλέπετε πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οποιουσδήποτε μπορεί να στείλει mail, σχόλιο, ακόμη και το ρεπορτάζ το δικό του. Και εμείς το δημοσιεύουμε. Εμείς χρησιμοποιούμε την Google Maps για τους χάρτες και μάλιστα έχω μια νέα εφαρμογή με ε, ειδικό χρωματισμό των συνοριογραμμών Οπότε έτσι βλέπουμε τα φυλάκια, βλέπουμε αν υπάρχουν σούπερ μάρκετ στα σύνορα, γενικώ οι λεπτομέρειε στα διάφορα σύνορα μεταξύ των χωρών. Αυτό το προβάλαμε και στην ιστοσελίδα μας. Και μάλιστα ε, θα ήθελα να αναφέρω εδώ τους εταίρους μας, Blog μία, ε, κάποιους φίλους ε, που μας στέλνουν από την Πολωνία και τη Γερμανία. Επίσης το Volo Blog που κάνουν τη γραμμή, την παλιά γραμμή Odernize, την έχουν διατρέξει με ποδήλατα. στάτ και ε, ένα πρακτορείο ταξιδίων που οργανώνει ταξίδια ακριβώ ε, και διαδρομές στα σύνορα. Όλοι αυτοί οι εταίροι μας είναι σημαντικοί γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έβλεπε το φως της ημέρας στο project μας. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα με το site αυτό. Το συζητήσαμε με τους ε, συναδέλφους ε, και χάρη στο βραβείο Σαλμάνια, Καρλομάγνου, θα, έχουμε, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το, την ιστοσελίδα μας, τον ιστοτοπό μας. Ε, θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στους επισκέπτες επίσης ε, του site μας, θα βλέπουμε ποιος επισκέπτεται. θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, θα διευρύνουμε το φάσμα των ρεπορτάζ, γιατί το επίκαιρο τώρα θέμα είναι η προσφυγική κρίση. Έχουμε συνεργασία και με τοπικές οργανώσεις, με την Oxfam, με μια γαλλική οργάνωση και θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τα ρεπορτάζ μας και προς αυτή την κατεύθυνση και θα συσφίξουμε τις σχέσεις και με τους εταίρους μας ε, ώστε να προβάλλουμε περισσότερο τον ιστοτοπό μας. Θα διαβρύνουμε και τη θεματολογία μας. Ε, για παράδειγμα, ε, θα κάνουμε μικρά ρεπορτάζ για τις εκλογές στη Γαλλία που θα γίνουν και στη Γερμανία το 2017. Θα έχουμε ένα παρατηρητήριο εκλογών. Θα αναλύουμε την κατάσταση, θα οργανώνουμε συζητήσεις Αυτά εν ολίγης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλο το επιτελείο της, του βραβείου Σαλαμάνια, του Καλομάγνου και κυρία την Άννη σατό για τις ωραίες εκδηλώσεις που οργάνωσε. Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη, τις πολύ καλές ιδέες, τις συζητήσεις και τις συναντήσεις που είχαμε στο Άχεν και τις Βρυξέλλες. Και αν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να απαντήσω. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και απλώς να σας πω το εξής. ναι, ναι. Di spegnere Σβήστε το μικρόφωνο. Απλώς να σας πω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ ε, αυτή η παρουσίαση για τα σύνορα που είναι κατά τόσο σημαντικό σήμερα. Συνάδελφοι, σας υπενθυμίζω ότι μια από αυτές τις ε, δημιουργίες ότι πρώτα-πρώτα αναλύθηκε από Επιτροπή Κριτική Εθνική, πρόσωποι του Κοινοβουλίου και κάποια φορά για τους νέους και κατόπιν έγινε μια δεύτερη διαλογή οπότε και προέκυψαν οι τρεις πρώτες. εκπρόσωποι του, του Ιδρύματος και τρεις βουλευτές. Κύριε Φρέμπ το πρέπει να φύγει, οπότε γι' αυτό και ζήτησε να μιλήσει. Πρώτα τώρα πάμε στο, τώρα πάμε τρίτο, στο τρίτο, Αυστρία. Soccer Social Club, Μιλώ. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μας δίνετε. Εγώ εκπροσωπώ την Αυστρία και το Social Soccer Club, αλλά επειδή μεγάλος θα μιλήσω γαλλικά. Ε, το Social Soccer Club τι είναι, είναι ένα τουρνά ποδοσφαίρου ε, και πάμε στην επόμενη διαφάνεια, κοινωνικού ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ και 13 χρόνια ο Ελμαρ Χάς, ε, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία στο Gratwein που είναι ένα χωριό δίπλα στο Grat της Αυστρίας. 5-6 νέοι λοιπόν τότε έφηβοι 15 χρονών σκέφτηκαν να αρχίσουν ένα πανευρωπαϊκό τουρνό ποδοσφαίρου. Και ο σκοπός ε, ήταν και απευθυνόταν σε νέους ηλικία 11 έως 18 ετών, αγόρια και κορίτσια. Είναι μεικτές οι ομάδες ποδοσφαιρικές, δηλαδή είναι υποχρεωμένες να έχουν τουλάχιστον ένα κορίτσι στην ομάδα τους για να μπορούν να συμμετέχουν λοιπόν ε, και κορίτσια στο τουρνουά ποδοσφαίρου. Κάθε χρόνο διεξάγεται αυτό ένα Σαββατοκύριακο τον Ιούνιο εδώ και 13 χρόνια. Στην επόμενη διαφάνεια είμαστε. Γιατί είναι ευρωπαϊκό αυτό το πρόγραμμα, διότι πάντα συμμετέχουν 20 ε, ομάδες, 100 ε, νέοι πάνω κάτω, οι περισσότερες ομάδες είναι ευρωπαϊκές, οι μισές και άλλες μισές είναι της εκάστοτε περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία μεταξύ των περιφερειών και της Ευρώπης γιατί θέλουμε να έχει και η Ευρώπη απήχηση στο τοπικό επίπεδο. Επίπεδο. Δηλαδή είναι φίλοι που μαζεύονται, κάνουν μια ομάδα ποδοσφαίρου 5x5 συνεργαζόμαστε και με τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια του χωριού κάθε φορά που διεξάγεται αυτό το τουρνουά για να υπάρχει και ε, βοήθεια στην τοπική οικονομία. Έρχονται οι ομάδες από τις υπόλοιπες χώρες. Τα 13 χρόνια που έχουμε αυτή τη διεξαγωγή του τουρνουά είναι 20 χώρες που έχουν συμμετάσχει. Ε, η Αυστρία είναι πάντα παρούσα και πολλές όμορες χώρες, ε, Ιταλία, Γερμανία, Ουγγαρία, συχνά προσπαθούμε να επεκτηνόμαστε και να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες. Εγώ φέτος δούλεψα για μια γαλλική ομάδα και η γαλλική πόλη Βιέν συμμετέχει. Ε, δεν είναι ε, πραγματικά ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, δεν είναι ομάδες νέων, είναι κοινωνικές ε, ομάδες από σχολεία, λύκεια, γυμνάσια. Δεν είναι αθλητική διοργάνωση, δεν είναι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Είναι φίλοι που έχουν κάνει μόνοι τους μια ομάδα ποδοσφαίρου τελείως ε, ψυχαγωγικού χαρακτήρα και όχι οργανωμένη σε αθλητικούς συλλόγους. Φυσικά ποδόσφαιρο είναι αλίμονο. Για το ποδόσφαιρο ε, κυριαρχεί όλο το Σαββατοκύριακο, ένα μικρό τουρνουά ε, που έχουν προκριματικές φάσεις και μετά τελική φάση τουρνουά κανονικό. Και είτε βγει πρώτη είτε τελευταία η ομάδα παίζει τον ίδιο ρυθμό αγώνων. Δηλαδή και τελευταίος να είσαι έχεις παίξει και τελικό παρηγοριάς και τέτοια αρκετά ε, σημαντικό αριθμό ε, αγώνων για να συναντιόνται οι ομάδες. Και δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό τουρνουά. Ακόμα και αν έρχονται οι νέοι για να παίξουν ποδόσφαιρο, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στο περιθώριο και στο πλαίσιο ε, του τουρνουά, παιχνίδια, κουίζ, θεάματα, συναυλίες, γεύματα, για να συναντιόνται οι νέοι και να ανταλλάσσουν απόψεις, να γίνονται φιλίες, να συζητούν για την Ευρώπη. Κάνουμε και μικρά εργαστήρια πολλές φορές που μπορούν οι νέοι να συζητούν για την Ευρώπη, τι, γιατί προσωπεύει για εκείνους η Ευρώπη. Δύο είναι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, δηλαδή κάθε φορά τέσσερι ομάδε μόνο παίζουν. Οι υπόλοιπε έχουν άλλε δραστηριότητε. Και με τον τρόπο του συμμετέχουν στην Ευρώπη. Πέσα πάντα στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού τουρνουά. Να βλέπετε εδώ φωτογραφίε από τα εργαστήρια που κάναμε τα τελευταία χρόνια. όπου οι νέοι περιγράφουν την Ευρώπη στη γλώσσα τους με τα δικά τους λόγια και στα αγγλικά. Είναι λοιπόν ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά Ευρωπαίων πολιτών. Και, αλλά όχι μόνο. Ε, συμβαίνουν διάφορα πράγματα, οι νέοι επικοινωνούν, γνωρίζονται. Και από αυτό το ποδοσφαιρικό τουρνουά που έχει ηλικία 13 ετών γεννήθηκαν πολλές φιλίες μια ομάδα από το Βέλιο και τη Γερμανία και έκτοτε κάθε χρόνο συμμετέχουν μαζί. Είναι ντόμινο, δηλαδή καταλήτης ε, αυτή η ε, διοργάνωση για πιο πολλές ε, γνωριμίες, φιλίες και επαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Grazie della vostra complimenti. Molti complimenti. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρος και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, διότι στην Ιταλία έχουμε κάτι ανάλογο για αυτό το κοινωνικό ποδόσφαιρο, ε, αλλά και αυτή η συμμετοχή σας για το ε, Κάρλο ε, παραπέμπει σε αυτές τις χώρες που έχουν μια τέτοια εμπειρία. Αλλά ξέρετε, είχαμε μια κρόαση και συζητήσαμε το πώς μέσα από αυτό αυτό το σπόρο όταν γίνεται σε τέτοιο, έχετε αυτή την κοινωνική διάσταση και μας οδηγεί σε καλύτερη κοινωνική ένταξη, σε φιλία, προσέγγιση, βοήθεια σε αυτούς που έχουν κάποιες δυσκολίες. Οπότε αυτό είναι η εφορμή το, το ποδόσφαιρο, αλλά τελικά οδηγεί σε καλύτερη κοινωνική ένταξη των νέων. Και τώρα... Πάμε στους νικητές το Λουξεμβούργο φέτος. Δεν είναι εδώ. Ah, sorry, sorry, no. Pensavo fosse fourth and, and five. Ah, no, no. The, the, the, the parity. Parity. Allora, tre premi, cioè tre... Ε... Επομένως, τρεις ήρθαν τρίτη. Οπότε, συμπάθημε κανένα Οπότε, έχουμε τώρα τη δεύτερη ομάδα που ήρθε τρίτη. Είναι η Κύπρος όσον αφορά το επιχειρηματικό πνεύμα ως λύση κατά της επασχόλησης. Ο Μάριος Αγαθοκλέος και ο Νικόλας Χριστοφή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσατε να έρθουμε για να σας παρουσιάσουμε το σχέδιό μας. Ο τίτλος είναι «Επιχειρηματικότητα, η λύση κατά της ανεργίας». Ξεκίνησε το 2014 από... και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νεολαία Ενδράση. Καταρχήν ποιοι είμαστε. Είμαστε ένα κέντρο νεότητας που ιδρύθηκε το 1998. Είμαστε μια εθελοντική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα ένα μικρό χωριό στην Ήπεθρο της Κύπρου. Είμαστε μια μικρή παρέα φίλων που προσπαθούμε να ψυχώσουμε τους νέους ε, να ε, ενταχθούν περισσότερα και πιο ενεργά στην κοινωνία. Και επίσης έχουμε μία μικρή λέσχη νέων. Θέλουμε, όπως σας είπα, να θερύνουμε τους νέους για πιο ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, να προωθήσουμε το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της νεολαίας της Κύπρου και γενικώ να φέρουμε τους νέους της Ευρώπης σε επαφή μεταξύ τους πώς ε, καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εναλλακτικές και καινοτόμες ιδέες τη επιχειρηματικότητα για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων στην Νότια Ευρώπη. Η μέθοδος μας ε, είναι μέσω της μη επίσημης εκπαίδευσης και μεθόδους μεθόδου ε, χρησιμοποιώντας χρησιμοποιώντα συστάσεις του πρώτου τρίου των Προεδριών της Ισπανίας, Βελγίου και Ουγγαρίας που ασχολήθηκε με το θέμα της ενεργείας των νέων. Εταίροι μας, το Κέντρο Νεότητας του Αγρού της Κύπρου, το ε, Youth Business Network από την Ελλάδα, η Ένωση Βαβέλα από, Βαβέλα από την Ιταλία, το Ραπλέξιον από την Κροατία και η υποστήριξη για την εξέλιξη των νέων της, της τελευταίας χώρας Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με οργανώσεις που έχουν παρόμοιες ε, με μας καταστάσεις, δηλαδή σε οργανώσεις από μικρά χωριά με υψηλό ποσοστό ανεργίας. Να σας παρουσιάσω τώρα τις μεθόδους που χρησιμοποίησαμε στο σχέδιό μας, στο project μας. Καταρχήν, ε, ζητούμε από τους συμμετέχοντες ε, να κάνουν μια αυταξιολόγηση των φιλοδοξιών τους, της εμπιστοσύνης τους, ε, της, των ηγετικών προσόντων που δείχνουν. Μετά ε, τους ζητούμε να χρησιμοποιήσουν την ε, καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Τους δίνουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν ένα σχέδιο δράσης. Επίσης δημιουργούμε πόστερα, φύσες και τους εφοδιάζουμε με υλικό που ίσως, θα, που ίσως το χρειαστούν και μετά παρουσιάζουν το υλικό τους σε ολιγομελές ακροατήριο. Μερικές από τις ιδέες που προέκυψαν από το σεμινάριο είναι ε, τα κούνη με ε, ύψος που μπορείς να το προσαρμόσεις. Επίσης, ε, μία διαφήμιση ε, μια εφαρμογή για να μπορεί κανείς να βρει θέση παρκαρίσματος, ένα gadget ε, πώς να βρει κανείς τα κλειδιά του που έχει χάσει, τον, το τον με τα κλειδιά του που έχει χάσει ή ένα spot τηλεοπτικό όπου μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μία εφαρμογή και να γράψει αυτά που θέλει και να βρει φίλους, ε, να βρει ε, ανθρώπους με κοινά με αυτόν ενδιαφέροντα. Επίσης, ε, εξετάσαμε το θέμα της ανεργίας ό,τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν είναι κανείς ε, άνεργος, είναι καταδικασμένος στο κοινωνικό αποκλεισμό. Γιατί εφόσον δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος, μένει στο σπίτι του, δεν έχει δουλειά, οπότε προτιμά να μένει μόνος, ε, κλεισμένος στο σπίτι και να μένει με σταυρωμένα χέρια. Ίσως χάνει και την αυτοπεποίθησή του και δεν έχει καν τη διάθεση να ψάξει για μια δουλειά. Οπότε προσπαθήσαμε να εξετάσουμε κάποιες πρακτικές για να καταπολεμήσουμε την, ε, την ανεργία. Και ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες τι προσπαθεί να κάνει κάθε χώρα κάθε κυβέρνηση στη χώρα τους για να καταπολεμήσει την ε, ανεργία. Μερικές φορές δίνει επιδόματα ή σύντομες εξάμηνες ε, θέσεις. Άλλοι έχουν μια τράπεζα ταλέντων όπου μπορεί κανείς να υποβάλει το βιογραφικό του και οι κρατικές αρχές υποτίθεται θα βρουν μια θέση, μια θέση απασχόλησης και προσπαθούμε να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις ε, συνέπειες της ανεργίας σε κάθε χώρα. Και μερικά από τα αποτελέσματα που επισήμαναν οι συμμετέχοντες είναι ότι οι καλύτερε πρακτικέ είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή γνώση και εμπειρίας για το θέμα της ανεργία των νέων, η, ανάπτυξη ενό ε, δημιουργικού και εφευρετικού επιχειρηματικού πνεύματος, η πρόθεση της συνεργασίας ε, ε, για το θέμα αυτό, η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσόντων και ε, μέσων για ένταξη στην αγορά εργασία και επίσης πρόθεση τη σημασία της κινητικότητας ε, για την προσωπική ανάπτυξη. Επίσης παρατηρούμε του νέους να βρουν τρόπους για να γίνουν πιο καινοτόμοι και πιο δημιουργικοί και εφάνταστοι. Γιατί η ιδέα είναι, αν δεν μπορείς να βρεις δουλειά, την εσύ, δημιούργησε εσύ μία θέση εργασίας. Ε, προσπαθούμε να αναλύσουμε και τις ε, ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους για να βρουν δουλειά. Το Erasmus ΣΥΝ, για παράδειγμα, το πρόγραμμα ή το Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες, το Eures Jobs, η εγγύηση για τους νέους, η πρωτοβουλία για τις ευκαιρίες της νεολαίας. Κάποιος από την Κροατία μίλησε για το Angels Den. Κάποιος ε, εύπορος χρηματοδοτεί καινοτόμες ιδέες που κρίνει χρήσιμες ε, και δίνει την ευκαιρία σε νέους να τις εφαρμόσουν. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, just, just... Ε, ευχαριστούμε και συγχαρητήρια τώρα. Πριν γίνουμε την τόσο σημαντική έκθεση όσον αφορά αυτές τις δεξιότητες για καταπολέμηση της ενδίας των εναυτών, αυτό εγκρίναμε. Και τώρα προχωρούμε. Ισπανία. Η Ισπανία πρόκειται να παρουσιάσει μια δημιουργία που ονομάζεται Info Actualidad. Δύο είναι οι δημιουργοί, η Κριστίνα Λονσογκαρσία και ο Χόρχε Κανιαβέρας. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, καλημέρα Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε πρώτα πρώτα το θα σας πούμε ότι το Infactorda είναι ένα ιντερνετικό περιοδικό που έχει ενημερωτικό ρόλο στα πλαίσια του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης γιατί είναι περίοδο ότι δεν υπάρχει στο Πανεπιστημίο αυτό ένα αντίστοιχο περιοδικό. Ε, ξεκινήσαμε το 2012 η κυρία Κάνερο ε, μας βοήθησε, μια καθηγήτρια και είπαμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην περιοριστούμε μέσα στους τοίχους του Πανεπιστημίου ή στα σύνορα της Ισπανίας, της Μαδρίτης. Θα πρέπει να έχουμε εμβέλεια πανευρωπαϊκή. Οπότε γι' αυτό έχουμε βάλει αυτό τον τίτλο, μια έκκληση προς την Ευρώπη, φωνή προς την Ευρώπη και έχουμε και διάφορους ε, ανταποκριτές ε, οι οποίοι συμμετέχουν στο έρασμος, να το πει την επόμενη διαφάνεια. Να που δεν τα πάει καλά. Λοιπόν, και είδατε ότι συμμετέχουμε σε πάνω από 30 πόλεις αυτή την τριετία και έχουμε 60 ανταποκριτές 25 προσθέτει κάθε χρόνο. Οπότε τι είναι αυτό, είναι μια σχολή για πρακτική. Μισό λεπτό, πετύχαμε ακόμα. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια διόρθωση. Γράφουμε ένα άρθρο, το διορθώνεται πριν δημοσιοποιηθεί, οπότε όπως γίνεται σε κάθε περιοδικό. Μια εφημερίδα ας πούμε. Και... Μισό λεπτό. Έχουμε το πρόβλημα με τις Βλέπετε το, τον χάρτη με τους ανταποκριτές μας σε όλες αυτές τις πόλεις. Από την Ελλάδα μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Βλέπετε τώρα ποια είναι η βάση αυτή τη δημιουργία, είναι οι ανταποκριτέ. Και όπω σας έλεγα, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει επομένω να έχουμε άμεση εποπτεία του τι γίνεται στι χώρε και πληροφορούμε για οι ειδήσει. Μπορείτε δείτε εδώ πέρα η εγκαθίδρυση του, του Πάπα Φραγκίσκου, ο, ο του Πρωθυπουργού Θάτσερ, αλλά και κάποια άλλα θέματα που τα μεγάλα ΜΜΕ δεν τα λένε. Ας πούμε μια συνέντευξη ενός ε, φρουρού Ελβετού ε, Μουσολίνη στη Ρώμη και είπαμε ότι βλέπουμε πόσα να έχουμε οι Ευρωπαίοι, τα οποία τα γνωρίζουμε και έτσι νομίζω ότι αναδεικνύεται αυτή η αίσθηση του είμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλο. Όταν πήγαμε στο Εράσμος είπαμε τι θα κάνω, φεύγω, πάω στις Βρυξέλλες και πώς λειτουργούν οι μεταφορές Φερρυπίν στις Βρυξέλλες. Οπότε μας τα λένε οι ανταποκριτές μας που μπορούμε να ψωνίσουμε, που είναι πιο φτηνά, που μπορεί να βγει κανείς να διασκεδάσει στην Ρώμη, πώς κανείς μπορεί από το αεροδρόμιο του Παρισιού να πάει στο κέντρο, επομένως, ο οδηγός επιβίωσης. Οπότε είπαμε θα πάμε να φοιτήσουμε, αλλά κάνουμε αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη. Άρα, πώς θα ταξιδέψει κανείς, ας πούμε, από το Παρίσι στις Βρυξέλλες για ένα ευρώ. Γιατί έτσι μαθαίνει κανείς τον κόσμο και έτσι κανείς αισθάνεται πιο Ευρωπαίος. Επίσης, κάνουμε και κάποια άλλα αμερόληπτα ρεπορτάζ. Δεν είναι όλα ρόδινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει μένως να βρίσκουμε και ποια είναι τα στραβά και τι κάνουμε, πάμε και συναντάμε κάποια κομμάτια του πληθυσμού, τμήματα του πληθυσμού, ας πούμε κάποιους παλαιούς φοιτητές, καθηγητές. Ε, ας πούμε βρήκαμε και τον κύριο Σέκα τον επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Ισπανία. Eurotrip. Συγγνώμη που δεν καταφέρνω με τα slides. Πιέζει και ο χρόνο. Ε, μετά το Eurotrip. Πού είναι αυτό. Α. Αυτό το οποίο βλέπετε τώρα αφορά το 75η επέτειο του, της λήξης του πολέμου. Έχουμε επομένω άρθρα από κάθε χώρα που γράφηκαν σε κάθε χώρα αυτό το αφιέρωμα ήταν αυτός ο λεθοσκοπευτής της Φιλανδίας ή μετά ήταν ο Χασάπης της Πράγας και δεν κάνουμε μόνο ρεπορτάζ αλλά επισυνεργαζόμαστε και με άλλους ε, κλάδους, άλλες σχολές του πανεπιστήμιου μας και έτσι έχουμε 9 πανεπιστήμια από 7 χώρες που ήρθαν στη Μαδρίτη για να τους εξηγήσουμε το πώς γίνεται αυτή η κοινωνική δουλειά στη Μαδρίτη Και βλέπουμε τα διάφορα κοινωνικά κινήματα, τι έχει γίνει στην Ισπανία, αυτά τα κινήματα με αφορμή την οικονομική κρίση και έτσι ήρθαμε σε επαφή και με άλλους Ευρωπαίους και τους είπαμε πώς δουλεύουμε στην Ισπανία, πώς μπορούμε να συντονιστούμε περισσότερο ο ένας με τον άλλο και ουσιαστικά αυτό είναι μια ανάσχεση στον ευρωσκεπτικισμό. Πάντως ότι δεν, αρκεί να μιλάει κανείς για την κρίση στην Ευρώπη, για την λιτότητα, για τις ε, Βρυξέλλες, αυτή η κακή ευρωβουλευτέ, όχι, θα πρέπει να δούμε το καλό πρόσωπο τη Ευρώπη επίση, ε, ολοκλήρωση, ο κοινό χώρο, η ΚΑΠ, όλα αυτά τα οποία δεν απασχολούν τα μεγάλα ΜΜΕ. Αυτό θέλουμε να προβάλλουμε. Οπότε είπαμε ότι η δημιουργία μας είναι κατά του ευρωσκεπτικισμού. Δεν λέμε ότι είναι όλα καλά και άγιοι ότι κάνουν Βρυξέλλε, αλλά ενημερώνουμε, ούτως ώστε οι νέοι στην Ευρώπη να μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη, το μέλλον μας. Το μέλλον μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, να συνεχίσουμε την ενημέρωση για την Ευρώπη από την Ευρώπη και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και feedback, κάποια ανταπόκριση αυτοί που στο έρασμος έρχονται στη, στο Μεσκήνα και βλέπουν τι γίνεται στην Ισπανία, πώς, τι γίνεται στη Μαδρίτη, άρα έχουμε συνέχεια κάποια ανταλλαγή, ανταλλαγή με την ευρωπαϊκή νοοτροπία, ούτω ώστε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν είμαστε από τη Μαδρίτη δεν είμαστε μόνο Ισπανοί, αλλά είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και συμπαθάτε με, λέει ο κύριο Κανιαβέρας, για τα προβλήματα τη διαφάνεια. Συγχαρητήρια, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε το πρώτο το οποίο θα κάνουμε είναι να δούμε αυτόν τον σύνδεσμο, ε, αυτό το link για να δούμε πώς προβάλλεται αυτό το πω ζουν οι νέοι. Πολύ ωραίο αυτό το δημιούργημα. Ε, και δώσουμε τώρα το λόγο στους νικητές του πρώτου, του Άνταμ και Λεγκέι, Λεγκάι, πώς ονομάζεται. Είναι το real time, WW1. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αυτά τα αρχικά τι σημαίνουν. Μπορούμε. Καταρχάς, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που έχουμε σήμερα, είμαστε εδώ. Οι δυο μας είμαστε από το Πανεπιστήμιο του ε, Λουξεμβούργου, μάστερ στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία και έχουμε έρθει να σας ε, παρουσιάσουμε αυτό το project. Ε, έχουμε εδώ ένα tweet που είναι ένα παράδειγμα των όσων κάναμε. Λέμε την ιστορία μέσα από το Twitter, την ιστορία του μεγάλου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τι έγινε με την ακριβή ώρα και την ακριβή ημερομηνία για το πώς το ζούσαν βασιλιάδες, κινηθνητοί, πρωθυπουργοί, ηγέτες ε, από ε, ένα ε, τραγούδι μέχρι την κήρυξη πολέμου από την Βουλγαρία στη Σερβία. Αυτό έγινε χτες, πριν από 100 χρόνια φυσικά. Το κάναμε αυτό για την εκατοστή επέτειο των Βαλκανικών πολέμων, έτσι ξεκίνησε και συνέχισε μέχρι την υπογραφή της συνθήκης των Βερσαλιών. Ε, είναι σημαντική η βοήθεια που είχαμε και θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα ε, από φοιτητέ από όλη την Ευρώπη που εργάστηκαν όλοι για το πρόγραμμα αυτό. Αυτό δείχνει ποιος είναι ο στόχος μας. Ε, να διηγηθούμε και πάλι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, όχι μόνο από την εθνική σκοπιά αλλά και την υπερεθνική. Και ο καθένας ε, έχει σημασία ανεξαρτήτως φύλου, προέλευση, κοινωνικής τάξης, καταγωγής κτλ ε, και κάποιοι followers στο Twitter μας θέλουν πληροφορίε, σχόλια κτλ. Είναι ένας λογαριασμός Twitter με tweet που έχουν γραφτεί σε καθημερινή βάση επαναλαμβάνω γεγονότα, προσωπικές ιστορίες, τι έγινε ακριβώς πριν 100 χρόνια, πριν από ένα αιώνα. Όλα τα tweet τα έχουν γράψει οι φοιτητέ στο Μάστερ Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Δημιουργούν νέε ιστορίες από το μεγάλο, το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και όσου το έζησαν. Κάθε tweet είναι μια φωνή ε, από το παρελθόν που φτάνει σήμερα σε όλους τους αναγνώστες και ακολουθητές στο Twitter. Και μέσω του Twitter ε, μοιραζόμαστε αυτό το ψηφιδωτό ιστοριών στα κοινωνικά δίκτυα. 10.000 μα ακολουθούν στο Twitter. Πάνω από 2.700 tweets έχουν ήδη δημοσιευθεί από το 2013. Κάθε μέρα τρία tweets βάζουμε. Αν και ο περιορισμός των 140 χαρακτήρων είναι πρόβλημα, ακριβώς αυτό μας ε, ε, προάγει να είμαστε δημιουργικοί. Αυτή η πλατφόρμα ε, είναι κάτι που ορισμένοι αμφισφητούν. Αλλά επειδή είμαστε φοιτητέ της ιστορίας, ε, συνδέουμε όλα τα tweet με ε, γνήσιες πηγές που έχουν ψηφιοποιηθεί για να βλέπουμε την προοπτική του καθενός ε, από την εθνική σκοπιά και την ευρωπαϊκή. Λοιπόν, για να δείξουμε ε, αυτό το πρόγραμμα έχουμε συνεργαστεί με πλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή τη Βιβλιοθήκη, με μουσεία για την εικονογράφηση. Εδώ βλέπετε ένα tweet που είναι ε, ένας πίνακα ζωγραφικής και τι κάναμε. Ε, ψάξαμε πάρα πολλά γράμματα, κάρτ ποστάλ, προσωπικούς λογαριασμούς, φωτογραφίες, γιατί ακριβώς εδώ είναι μαρτυρίες ε, όπως το έβλεπαν ε, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, αυτό το θέμα του πολέμου, για να μπορούν όσοι μας παρακολουθούν να δουν ε, και το πιο συναισθηματικό επίπεδο πέρα από το αμυγό ειδησιογραφικό. excuse me. Next Το επόμενο. Εδώ είναι μια κάρτα ποστάλ, προπαγάνδα βρετανική. Έχουμε παραδείγματα από όλο τον κόσμο τέτοια γερμανικά, ρωσικά, γαλλικά κτλ. Βασικά σε κάθε χώρα που συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τα ίδια μηνύματα για να εμψυχώνουν τον κόσμο να πολεμάει. Ανεξαρτήτως γλώσσας, ε, πολιτισμού, μεθόδου, η εμπειρία είναι η ίδια. Και δείχνουμε λοιπόν με αυτό το project ότι ακόμα και στη σύγκρουση έχουμε ομοιότητες ξεπερνάμε το εθνικό αφήγημα και δείχνουμε ότι υπάρχει ε, κάτι που ονομάζεται κοινή ευρωπαϊκή ιστορία. Εδώ βλέπετε ένα θάμνο που περπατάει. Είναι ένας Τούρκος ελεύθερος σκοπευτής με, σκοπευτής που μόλις έχει ε, πιαστεί εχμάλωτος. Αυτό είναι ενδιαφέρον βλέπουμε κάποιες ιστορίες που έχουν χαθεί. Το 1917 ένας Γάλλος, τρελή ιστορία, προσπάθησε να καμουφλάρει το Παρίσι ολόκληρο ε, για να έρχονται τα Ζέπελιν, τα αερόστατα αυτά και να βομβαρδίζουν λάθος πόλη. Ε, αυτό προφανώς απέτυχε, αλλά έχει ε, χαθεί και από την κοινή γνώση. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Αυτές τις χαμένες ιστορίες θέλουμε να τις επαναφέρουμε ε, στη ζωή και στην επικαιρότητα. Επόμενη διαφάνεια. Το σχέδιο μας λοιπόν θέλει να δείξει κάθε πτυχή του ε, πολέμου και δίνουμε σε όσους μας παρακολουθούν την πραγματική ζωή τι συνέβαινε ακριβώς πριν από 100 χρόνια. Φέρνουμε ε, την ιστορία στο παρόν και δείχνουμε την κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα, οι Γερμανίδες, οι αυστριακές γυναίκες δεν μπορούσαν ε, να φτιάξουν γλυκά γιατί η τιμή της ζάχαρη είχε εκτοξευτεί ας πούμε ή δεν βρίσκανε αλεύρι. Οπότε ε, άλλαξε ο πόλεμος στην καθημερινότητα και στα πιο μικρά πράγματα και πέρα από το εκπαιδευτικό και το ενημερωτικό του προγράμματος αυτού είναι τι σημαίνει να ζει σε μια διαιρεμένη Ευρώπη πριν από 100 χρόνια για να καταλάβουμε ακριβώς τι εστί να ζούμε σήμερα σε ειρήνη στην Ευρώπη αυτή. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια πολλά. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δέσμευση και την προσήλωσή σας και το βλέπουμε μέσα από τα μάτια των νέων, των σημερινών αυτό το παρελθόν και τη συναισθηματική προσέγγιση αλλά και την αυστηρή επιστημονική και ιστορική προσέγγιση. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. χρησιμοποιείτε το Twitter ε, με αυτόν τον τρόπο και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος καινοτόμο τρόπος. Ελπίζω να το συνεχίσετε. Μέχρι το 18 προφανώς που τελειώνει ο πόλεμος. Ε, και θα τελειώσει το project αυτό, αλλά είμαι βέβαια ότι θα συνεχίσετε, γιατί και με πάθος εργάζεται και με αποφασιστικότητα. Πριν δώσουμε τον λόγο στους ανθρώπους που έχουν ζητήσει τον λόγο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ε, σήμερα έχουμε την εξή ρύθμιση. Έχουμε πρώτα-πρώτα ε, αυτή την έκθεση που ψηφίσαμε όσον αφορά τις δεξιότητε που χρειάζονται για την ανεργία των νέων και επίσης σήμερα θα μιλήσουμε ε, και για κάποια έκθεση που έχει θέμα το πώς θα διδάσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία. Οπότε είστε ότι πρέπει για να προωθηθεί αυτό το θέμα. Και η τρίτη σημαντική έκθεση που σήμερα θα συζητήσουμε είναι η έκθεση Word όσον αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις ε, εκπαιδευτικές προκλήσεις. Έχετε πολλά να μας μάθετε σε αυτό το επίπεδο. Η Πέτρα Κάμερβερτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους ε, τους βραβευθέντες που έχουμε εδώ σήμερα. Είναι καταπληκτική η δουλειά πραγματικά που έχετε κάνει και ελπίζω να συνεχίσετε και στο μέλλον. Μπορώ να φανταστώ πάρα πολύ καλά ποιες δυσκολίε αντιμετώπισε η Κριτική Επιτροπή για να κρατήσει μία σειρά και στα βραβεία. Και επίσης φέτο το γεγονό ότι έχουν ισοβαθμίσει τρεις στην τρίτη θέση είναι πάρα πολύ εύγλωτο και δείχνει πόσο δύσκολη ήταν η επιλογή της Κριτικής Επιτροπής. Κάθε project που ακούσαμε σήμερα το πρωί είναι καταπληκτικό, μεγαλειώδες, καλύπτουν όλα αυτά διάφορους τομείς, αλλά κυρίως μας δείχνουν ότι όσα προβλήματα και να έχουμε σήμερα, όσες προκλήσεις και να αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, όσο ευρωσκεπτικισμό και αν βλέπουμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι από κοινού με άλλους νέους από άλλα κράτη-μέλη, αλλά και πέραν αυτών θέλουν να συνεργαστούν έτσι ώστε η Ευρώπη μας να γίνει καλύτερη, να αξίζει να ζει σε αυτή και να διατηρηθεί στο μέλλον. Και ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο παράδειγμα, να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, ε, σε μια κατάσταση που έζησε η Ευρώπη, ο πόλεμος που δημιούργησε πάρα πολλά δεινά και πολύ μεγάλο πόνο προκάλεσε έχει σημασία να δείχνουμε ότι αυτό δεν αφορά τη μεγάλη ιστορία των κρατών, αλλά και τη μικρή, τις μικρές καθημερινές ανθρώπινες ιστορίες. Τι σημαίνει να ζεις ένα πόλεμο. Γιατί τα τελευταία 70 χρόνια δεν το έχουμε ζήσει και το έχουμε επιτύχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να φανταστεί, φαντάζομαι, τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνει στα σύνορα, να δείχνει διαβατήριο και να μην σε αφήνουν καμιά φορά να περνά και τα σύνορα. Δηλαδή να μην επιτρέπεται να φορά γαλλικά ρούχα, ας πούμε, γιατί είναι ο προαιώνιο εχθρό. Σήμερα είναι όλα αυτά τόσο προφανή και αυτονόητα που δεν μα περνάνε από το μυαλό καθόλου. Καλό είναι λοιπόν να γυρνάμε καμιά φορά τα μάτια μας στο παρελθόν και να βλέπουμε τι έχουμε επιτύχει αλλά και να στρεφόμαστε και προς το μέλλον για να δούμε τι μας απομένει να κάνουμε. Γι' αυτό ε, αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας ε, των νέων, όπως το project που ακούσαμε από την Κύπρο, και να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ε, να δημιουργήσουν οι ίδιοι δουλειέ για να βγουν από αυτή την κατάσταση, να αναρωτηθούν τι μπορώ να κάνω εγώ για να βγω από την ανεργία και όχι να περιμένω πάντα από κάποιου άλλου να με βγάλουν. Πολύ ωραία, καταπληκτικά όλα αυτά τα project λοιπόν και το θέμα του Εράσμους αυτό το πρόγραμμα Erasmus Plus είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχής που καταφέραμε να το συνεχίσουμε. Και επίσης επιτύχαμε έστω και μικρή αύξηση των κονδυλίων για την τρέχουσα περίοδο. Γιατί ακριβώς αυτή η ανταλλαγή των νέων ε, σημαίνει το μέλλον της Ευρώπης. Κάποιος μίλησε για ντόμινο. Είναι γεγονός αυτό. Ελπίζω να επεκταθεί και πέρα από όλα αυτά τα σχέδια τα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Είναι καταπληκτική η δουλειά που κάνετε, ο ενθουσιασμός, η προσήλωσή σας και παρακαλώ να μην χαλαρώσετε. Και όταν τα βλέπω όλα αυτά, ομολογώ ότι δεν φοβάμαι για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, συμφωνώ με όλα αυτά όσα είπα και τώρα το λόγο η Τζούλι Ward και κατόπιν η Τρούπελ Ward. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα παρουσιάσω και εγώ την έκθεσή μου, αλλά θα ήθελα να πω πόσο, πόση χαρά νιώθω. Πραγματικά είμαι έμπλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη, είμαι από την Νοτιοδυτική Αγγλία, αλλά αισθάνομαι πραγματικά Ευρωπαία και βλέπω πόσο ελπιδοφόρο είναι το έργο της νεολαίας. Χθες είχαμε και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Βραβείου Πολιτών και ο Τζάφα είναι πίσω και πραγματικά κέρδισε χθες το βραβείο ε, μας εμπνέει πολύ το έργο του, το ίδιο και το δικό σας. Και αυτό το δίκτυο που επιτρέπει στους νέους να έρθουν πιο κοντά, ακυρώνει ουσιαστικά τα σύνορα και φέρνει κοντά τους νέους γύρω από ένα κοινό προβληματισμό, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης γίνεται και μία κριτική ανάλυση του θέματος και ελπίζω να φτάσουν μέχρι και τη δική μου πατρίδα τα project σας. Έχουμε πρόβλημα με το νερό, γιατί είμαστε νησί και μερικές φορές έχουμε περισσότερους δεσμούς με την υπηρετική Ευρώπη από ό,τι μεταξύ μας ε, στη χώρα. Και τέτοιου είδους προγράμματα πραγματικά γεφυρώνουν αυτό το ε, χάσμα, αυτό το νερό, το υδάτινο στοιχείο που μας χωρίζει. Και ο Τζάφα πραγματικά επιτελεί επίση εξαιρετικό και αξιέπαινο έργο στον τομέα του. Μερικές φορές ούτε εμείς οι ευρωβουλευτές δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση ε, και να κινηθούμε μέσα στην Ευρώπη. <laughs> Ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε την εφαρμογή και το σχέδιο που μας παρουσιάσατε για να κυκλοφορήσουμε να βρούμε θέση στάθμευσης στην Ευρώπη. Γιατί πραγματικά σήμερα το πρωί είχα προσωπική εμπειρία πόσο δύσκολο είναι. Όντω ε, θα μα βοηθήσουν τέτοιες σχέδια. Κυρία Τρίπελ, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις γιατί δείχνεται πραγματικά ζήλο, ζέση, ενθουσιασμό και στράτευση ε, για, στην, ε, για την Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρώπης. Πολύ ζωηρό ενδιαφέρον εγείρει λοιπόν ε, αυτό το, αυτό το σχέδιο γιατί δείχνουν πραγματικά δείχνει ευρωπαϊκές ιστορίες, ευρωπαϊκά βιώματα και περιπτώσεις τέτοιες ευρωπαϊκής προσήλωσης και χαίρομαι γιατί το βραβείο Καρλομάγνο σας έδωσε την ευκαιρία να συναντήσετε άλλους νέους και να ανταλλάξετε μεταξύ σας απόψεις. Πολύ σημαντική λοιπόν η συνεισφορά αυτή και χαίρομαι που βλέπουμε πραγματικά τους ε, καρπούς και τα ωφέλη αυτού του βραβείου. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο το ιστορικό των ε, σχεδίων σας. Από πότε τα ξεκινήσατε και πώς αποφασίσατε να υποβάλλετε συμμετοχή για το βραβείο Καρλομάγνος. Υπήρχαν ήδη άλλα σχέδια που σας ενέπνευσαν. Μπορείτε να μας πείτε λίγο το ιστορικό πώς καταλήξατε στο project σας και την υποψηφιότητα για το βραβείο Καρλομάγνος. Ποιος θέλει να απαντήσει σε αυτές τις ε, ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι έγινε με αυτά που φτιάξατε. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δώσετε κάποια συνέχεια σε αυτά που κάνατε. Έχετε το λόγο. Okay. Ε, ε. Για το ισπανικό project, εμείς πώς ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 12 και ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θέλαμε να απευθύνουμε μια έκκληση στην Ευρώπη και να ενημερώσουμε για την Ευρώπη. Αναγνωρίζω ότι δεν είχαμε ιδέα ότι υπήρχε το βραβείο Καρλομάγνους και τέτοια. Τίποτα, καμία σχέση. Ε, θέλαμε απλώς ε, ως δημοσιογράφοι να δράσουμε για την εφημερίδα μας και επειδή ε, αισθανόμαστε Ευρωπαίοι και η ηλεκτρονική εφημερίδα είναι ένα σχέδιο στραμμένο προς το μέλλον. Κάθε χρόνο βελτιώνουμε το δίκτυο, την ομάδα, τη διευρύνουμε. Είμαστε 140-400 φοιτητές δημοσιογραφίας πέρασαν από το περιοδικό μας τα τρία χρόνια, από την εφημερίδα αυτή την ηλεκτρονική και ε, το συζητούσα με τη Χριστίνα εδώ, τη συνάδελφό μου. Και μας είπαν «Ε, είστε σε καλό δρόμο και τα λοιπά, αλλά προσοχή υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα. Γιατί ακόμα πολλοί επικρίνουν την Ευρώπη και θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές ε, αποφάσεις είναι λαθασμένες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Άλλος, άλλη. Ναι, σε ό,τι αφορά το γαλλικό, ε, το, το αυστριακό, το ποδοσφαιρικό τουρνουά, 13 χρόνια είπαμε, ε, το έχουμε και το βραβείο Καρλομάγνου ήταν κάπως ουρανοκατέβατο και ξαφνικό. Ψάχναμε στο διαδίκτυο και είδαμε, α, κοίτα τι υπάρχει, βραβείο Καρλομάγνου. Και ομολογώ ότι τον συνειδητοποιήσαμε εκ των υστέρων. Εμείς τι κάναμε, ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά και ξαφνικά καταλάβαμε ότι κοίτα, έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Εγώ δεν είμαι όλα αυτά τα χρόνια, 13 χρόνια, αλλά οι άλλοι συνάδελφοι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ούτε εγώ τι επιπτώσεις και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ένα τέτοιο project και απευθυνθήκαμε σε αυτό το βραβείο που μας αναγνώρισε τη δουλειά που κάνουμε και πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πάρα πολύ. Είναι μεγάλη ικανοποίηση. Κοιτάξτε, το 2013 στο Λουξεμβούργο θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση για τα 100 χρόνια ε, του πολέμου, την επέτειο. Αυτό ακυρώθηκε όμως, το ακύρωσε η κυβέρνηση. Εμείς ως ιστορικοί όμως αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα δικό μας project και το 2013 αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε τι να κάνουμε ε, και πώς να το παρουσιάσουμε. Ουσιαστικά πριν το βραβείο Κάρλο Μάγνου γνωρίσαμε μεγάλη καχυποψία, αντιστάσεις, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τι θέλετε τώρα τόσα χρόνια πίσω, ένα αιώνα πριν. Όταν όμως κερδίσαμε το βραβείο Καρλομάγνου, ε, μας δώσανε προσοχή στο Λουξεμβούργο και περισσότερους ε, followers είχαμε στο Twitter, γιατί ουσιαστικά οι περισσότεροι followers είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Και η Ευρώπη ήταν όψιμη η κατάκτηση μετά το βραβείο. Μας βοήθησε λοιπόν να έχουμε followers. Η ιδέα προέκυψε από τι ανάγκε των νέων τη ε, κοινότητα και τη Κύπρου γενικότερα. Ε, πούμε ότι δραστηριοποιούμαστε σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα τελευταία έξι χρόνια. Ε, κάναμε περισσότερα από 25 προγράμματα ε, βάσει των αναγκών πάντα των νέων. Ε, Βλέποντα ότι η ανεργία των νέων είναι νούμερο ένα ε, πρόβλημα στην Ευρώπη, ε, είπαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Ε, βρήκαμε συνεργάτε αξιόπιστους ε, του οποίου συνεργαζόμασταν ε, και πιο παλιά και είχαμε επίση τα αποτελέσματα από την τροπολετρία που είχε να κάνει σχετικά με την εργασία των νέων, άρα αξιοποιήσαμε αυτά τα, τα στοιχεία. Για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνο είμαστε γνωστέ, γιατί συμμετείχαμε από το 2010 και σε εθνικό επίπεδο κατακτήσαμε το βραβείο το 2010 και 2011. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Allora, Πριν di tutto, Και πάλι συγχαρητήρια και ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ο Βασιλιακής δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχίσουμε την επαφή μαζί σα. Και πολλές φορές ε, απονέμεται ένα βραβείο, δεν δίνεται συνέχεια. Οπότε ε, είπαμε ότι θα υπάρχει μετάδοση στο ίντερνετ και να παρακολουθήσουμε το τι θα γίνει. Ε, όποτε έχετε κάτι να μας ε, πείτε, να μας προτείνετε, είμαστε ανοιχτοί. Οπότε σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για τη βοήθεια και τον Ιτίν Φράνσις Γκούτμαν μια που ήταν τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η ομπειρία και για την υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Γιατί ακριβώς θα πρέπει και οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου να ευαισθητοποιούνται και να ευαισθητοποιήσουν για μια που δεν είναι τόσο γνωστό αυτό το βραβείο. Να το ξέρουν καλύτερα οι ΝΟΕ. Και επίσης να ε, μάθει και ο κόσμος ποιοι πήραν τα βραβεία. Γεια σας. solo un momento Bene, allora. Πρόεδρος. Ωραία. Και τώρα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων. Έκθεση Δράγκητσα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Αφορά την διδασκαλία ή το μαθαίνοντας, μαθαίνοντας το σχολείο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούσαμε τους ε, νέους, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον, οπότε είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει επαφή με τις οργανώσεις των νέων, να δούμε τι θέλουν, τι, ζητάνε, τι προτείνουν. 12 Νοεμβρίου θα γίνει η επόμενη συνάντηση για να συζητηθεί η έκθεση και στις 11 πρώτου του 16 θα γίνει η ψήφιση. Ε, συνάδελφε Ντράγκητς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία για σύνταξη έκθεση με αυτό το θέμα, μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχόλια. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, ιδιαίτερα στο, στο τωρινό πλαίσιο, τώρα που αντιμετωπίζουμε τόσο σημαντικές προκλήσεις. Έξαρση του ευρωσκεπτικισμού, κάτι που θα ε, πλήξει την Ευρώπη και θα υπονομεύσει τις ε, θεμελιώδεις αρχές. Επίσης έχουμε έξαρση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ε, καταστρατήγηση της δημοκρατίας από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, ε, ένα χάσμα και μια μεγάλη απόσταση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών, γιατί κατηγορείται για έλλειψη δημοκρατικού ελλείμματος η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες και ότι στρέφει την πλάτη στους πολίτες ε, χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογές και περιορισμένη γνώση στο ευρύ κοινό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη ε, και οι νέοι δεν γνωρίζουν ε, τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και ανησυχητικό. Για παράδειγμα, το 2014, ε, σφιγμομέτρηση του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι 71% των Ευρωπαίων πολιτών νιώθουν ότι δεν είναι καλά ενημερωμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 44% αισθάνονται ότι δεν καταλαβαίνουν αρκετά πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτές λοιπόν τις ε, περιστάσεις ε, δεν ε, μας ξενίζει η αλωτρίωση που αισθάνονται και η απόσταση που αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες από το ευρωπαϊκό σχέδιο και το ευρωπαϊκό όραμα και ότι αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός και η επίκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοκρατικό έλλειμμα στις διαδικασίες. Ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν νιώθουν ότι συμμετέχουν στο δημοκρατικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταλαβαίνουν τι έγινε με τις ευρωεκλογές. Μόνο 27% των πολιτών, ε, ε, των νέων, και κάτω από το 40 των πολιτών ψήφισαν. Υπήρχε μεγάλη αποχή λοιπόν από τις εκλογές. Ήταν η χαμηλότερη προσέλευση στις κάλπες από το 1979, την πρώτη άμεση καθολική ψηφοφορία. Οπότε θεωρώ ότι αν ενημερώσουμε καλύτερα του πολίτες ε, θα ενθαρρυνθούν για να συμμετέχουν καλύτερα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι στόχοι μας ε, που ε, έχουν να, να προετοιμάσουν τον κόσμο για την εκπαίδευση και να τους καταστήσουν ενεργούς πολίτες. Επίσης να συνδέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους πολίτες. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο υπήρχε στο πρόγραμμα των πολιτικών από το 1976. Τότε είχαμε το πρώτο πρόγραμμα στην παιδεία. Είχαμε και το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας το Φεβρουάριο του 1976 και ένα πρόγραμμα δράσης για την παιδεία. Με την υιοθέτηση των 92 της συνθήκης του Μάστριχτ ε, προέκυψε και νομική βάση για την ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην παιδεία. 149 το, στο Μάστριχ, 165 τις συνθήκες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, μπορούμε να προαγάγουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να προωθήσουμε τις, την εκμάθηση των γλωσσών ή την κινητικότητα των διδασκάλων και των φοιτητών, των σπουδαστών ή να προωθήσουμε ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις βέλτιστες πρακτικές ή να προωθήσουμε ανταλλαγές ε, φοιτητών και καθηγητών. Από το πρόγραμμα δράση του 1976 πολλά ψηφίσματα και προγράμματα έχουν υιοθετηθεί και πολλές πρωτοβουλίες έχουν εγκριθεί για να προωθήσουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία και στα πλαίσια τη στρατηγική του 2020. Και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση για τους νέους 2010-2018 ε, και πρόσφατα η διακήρυξη των Παρισίων του Μαρτίου του 2015 των Υπουργών Παιδεία, αλλά και το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 για την εφαρμογή του Erasmus Plus και τη δέσμευση για να δώσει σάρκα και οστά στη διακήρυξη των ε, Παρισίων έφερε, την, ε, με δυναμικό τρόπο τη διάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παιδεία. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα ε, διευρυμένα και να προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους πολίτες. Εμείς βέβαια επικεντρωνόμαστε σε μία πτυχή, το πώς θα μάθουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα την προωθήσουμε μέσω της εκπαίδευσης. Γιατί η σχολική κατάρτιση θα πρέπει να εφοδιάσει τους σπουδαστέ ε, με γνώσεις για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις ε, θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και το πώς θα επηρεάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την καθημερινότητα και την ε, πατρίδα τους. Έτσι θα τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν για να γίνουν ενεργοί πολίτες και στην Ευρώπη και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Τώρα, ποιες είναι οι εθνικές προκλήσεις. Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει συμπεριλάβει την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχολικά προγράμματα και στις επιμορφώσεις και καταρτήσεις των καθηγητών. Υπάρχουν όμως διαφορές και εντός των κρατών μέλων, στο εσωτερικό τους και μεταξύ των κρατών μέλων. Οπότε πολλά θα πρέπει να κάνουμε ακόμη. Για τα σχολικά προγράμματα, επιμόρφωση των καθηγητών, εγχειρίδια σχολικά ή μέθοδοι διδασκαλίας, γιατί μερικε φορές είναι πολύ γενική προσέγγιση που υιοθετείται ή πολύ κατακαιρματισμένη. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη συνοχή και συμπληρωματικότητα με το υπόλοιπο σχολικό υλικό. Ή δεν είναι επαρκώ καταρτισμένοι οι καθηγητέ, οι δάσκαλοι για να διδάσκουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η επιμόρφωση. Επίση, τα σχολικά εγχειρίδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη κάλυψη των ε, κοινοτικών θεμάτων και να προσαρμόζονται στις διάφορες ηλικιακέ ομάδες και να λαμβάνουν υπόψη τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και σπουδαστών. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διαδραστικά μοντέλα διδασκαλίας ε, για να δίνονται ενάψματα στους ε, σπουδαστές ε, να εντρυφήσουν στο θέμα αυτό και να δουν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει και την καθημερινότητά τους. Έτσι θα αναπτύξουμε κοινωνικές δεξιότητες και θα προετοιμάσουμε τους συμπολίτες μας να γίνουν πραγματικά ενεργοί πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες επίσης δεξιότητες θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην επίσημη παιδεία, στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα και να δημιουργηθούν καλύτερη σύνδεση μεταξύ της επίσημης, ανεπίσημης και μη τυπικής ε, ε, διδασκαλίας. Με τέτοια προγράμματα όπως το Erasmus Plus ε, και το Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και τον διαπολιτισμικό ε, διάλογο και την διαπολιτισμική κατανόηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινητικότητα και ε, δαψιλή δημοσιονομική στήριξη, ώστε να έχουν όλα αυτά τα προγράμματα θετικά, θετικές συνέπειες για τους συμμετέχοντες και να έχουν ευρεία συμμετοχή. Οπότε χαιρετίζω το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 για την εφαρμογή του προγράμματος Erasmus Plus και τη δέσμευσή της ε, να δώσει συνέχεια στη διακήρυξη των Παρισίων. Κυρίως ε, στο να αυξήσει τον αντίκτυπο του Erasmus ε, στη δημιουργία της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, του πολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της ελληνικής και να στηρίξουν και τις οργανώσεις των πολιτών που έχουν σημαντικό ρόλο. Ε, τα θέματα της αδελφοποίησης πόλεων ε, και διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες ε, καθώς και κατάρτιση ενηλίκων συμβάλλουν σε αυτό το στόχο της καλύτερης εξοικείωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες εικονικές πλατφόρμες όπως το Teacher's Corners, η, γωνία του, η γωνιά του δασκάλου και του καθηγητή, δίνει πληροφορίες και υλικό για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διευκολύνει την πρόσβαση σε ενημερωμένο και επικαιροποιημένο διδακτικό υλικό. Τα υπάρχοντα δίκτυα προωθούν την εξοικείωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα και θα πρέπει να ενισχυθούν. Επίση, η ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών μεταξύ των δικτύων θα πρέπει να προωθηθούν. Έτσι, μπορούμε να προσεγγίσουμε την ηλεκτρονική μόρφωση ε, και υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία και να έχουμε συνεχείς επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινωνία των πολιτών. Και στο σεμινάριο ε, θα έχουμε και σχετικό σεμινάριο με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και περιμένω και τα σχόλια των συναδέλφων. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ φιλόδοξη και ολοκληρωμένη προσέγγιση σας και χαίρομαι που ε, αυτό το τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα ε, έχει όλες αυτές τις ε, πτυχές του διαπολιτικού διάλογου, της ε, εμπλοκής των πολιτών. Οπότε πρόκειται και εδώ για μια μεγάλη πρόκληση. Και οπότε πάρα πολύ ευχαριστώ το ότι σας απασχολεί με τόσο ενδιαφέρον. Και τώρα να μιλήσουν οι συνάδελφοι και κυρίως οι σκιώδεις ηγητές. Μάουρο έχει δει στο λόγο και κατόπιν οι υπόλοιποι έχουν δει στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω με την ε, σύντομη παρέμβασή μου από κάτι που είχε πει ο Ζωμονέ, ο οποίο, για τον ρόλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έλεγε εμείς ενώνουμε και φέρουμε κοντά τον κόσμο, όχι τα κράτη. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια ε, δυναμική εμπλοκή σε αυτή την ε, εκπαίδευση του ΣΥΠΗΝ. Οπότε να έχουμε αυτές τις γέφυρες και αυτό να πηγαίνει πάρα πέρα από τις εθνικές ε, ταυτότητες, τις κρατικές ταυτότητες. Οπότε έχουμε αυτά τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα για έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, τα οποία είναι προσανατολισμένα προ την επίτευξη αυτού του στόχου. Και επομένω με αυτή την αφετηρία που έχει και ε, μεθοδολογικό χαρακτήρα αλλά και διανοητικό, πνευματικό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, είναι κάτι το οποίο επήγει, να υπάρχει μια τέτοια συνειδητοποίηση και ταύτιση με την Ευρώπη, μια που η Ευρώπη τώρα ε, έχει πάρα πολύ δύσκολες προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει την σήμερα ημέρα. Για μια μεριά έχουμε την ανάδυση των λαϊκισμών και των εθνικισμών και βλέπουμε ότι θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της η Ευρώπη μακριά από, τη, από τα, στενά ε, συμφέροντα και οπότε ε, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε αυτούς που αμφισβητούν την ε, νοημοποίηση της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μια όθηση για να γίνει η Ευρώπη διεθνής παίκτη και πρωταγωνιστής στη διεθνή σκηνή και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει μέσα στην ύλη των πανεπιστημίων και θα πρέπει από το σχολείο να διδάσκονται οι επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω να λέω καλά το όνομα του κύριου Ντραγίτσα, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας έκανε και την ε, ε, εισήγησή του. Και ε, επίσης, ε, μπράβο που έχει τέτοια φιλοδοξία για το θέμα του. Οπότε ε, θα πρέπει να δάσκει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία όπως λέει η έκθεση οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αφετηρίας η Ευρωπαϊκή έχει κάνει μια μελέτη σχετικά και λέει ότι στην παιδεία ε, θα πρέπει να δάσκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ και πολλά χρόνια αυτό είναι στο θεματολόγιο της Ένωσης και νομίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να δώσει μια τέτοια όθηση για μια τέτοια παιδεία του κόσμου, ούτως ώστε τα σχολεία ε, και τα λοιπά τα ιδρύματα να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μάθουν την ε, σημασία ε, της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι μηχανισμοί των προστασίας των δικαιωμάτων όπως ενσωματώνται στις συνθήκες και επίσης για το ότι όλα αυτά είναι κοινέ αξίες, κοινέ αξίες πολλών εκατομμυρίων. Ευχαριστώ. Ή Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφε Μάουρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να αποδειχτώ συνεργάσιμο στην Επιτροπή αυτή και να δω και την προστιθέμενη αξία της σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά αμφισβητώ βαθύτατα την αξία αυτού του θέματος. Και ε, ο ευρωσκεπτικισμός και η ξεροφοβία συγχέεται με τον άκρατο εθνικισμό. Καμία σχέση και εδώ μέσα και στην Ευρώπη ε, ο κόσμος μπορεί να αμφιβάλλει για τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ ε, περιστατωμένο και στοιχετημένο σε πολλές φορές. Ακούω ότι θέλετε να διδάξετε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία, δηλαδή πόσο καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα και ο κίνδυνος της παρούσης έκθεσης η ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε για να μπορεί ο κόσμος να έχει κριτική σκέψη. Αλλά η προπαγάνδα για το πόσο σπουδαίο είναι το λεγόμενο ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι το τελείως αντίθετο και είναι και τελείως ε, ε, καταδικαστέο. Άκουσα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, για το σκεπτικισμό ότι είναι κακό και να μαθαίνουμε στον κόσμο να μην αμφιβάλλει. Αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα, είναι ύβρις προς τους πολίτες και τα δικαιώματά τους να αποφασίζουν μόνοι τους. Και ιδιαίτερα αμφισβητώ αυτή την παραδοχή ότι μαθαίνουν, όσο περισσότερα μαθαίνουν για την Ένωση οι πολίτες, τόσο περισσότερο τη λατρεύουν και οι ευρωσκεπτικιστές είναι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει πόσο φανταστικοί είμαστε και πόσο σπουδαία και ε, καταπληκτικά και μεγαλειώδη πράγματα κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, υπαγορεύει στα κράτη-μέλη τα προγράμματα σπουδών των σχολείων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν αγωγή του πολίτου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο διδάσκεται και τονίζεται και από τα δύο βασικότερα κόμματα ε, το να λένε τώρα οι ε, βουλευτές και Ευρώπη τι θα διδάσκουμε στα σχολεία είναι πραγματικά εξωφρενικό. Ε, Βεβαίω, βέλτιστε πρακτικέ και να διδάσκονται το ένα κράτο από τα άλλα, αλλά αυτά που άκουσα ε, δεν είναι καθόλου βέλτιστε πρακτικέ. Η Ευρώπη για του πολίτε δεν είναι καθόλου βέλτιστη πρακτική σε καμία περίπτωση. Και εγώ έχω καταθορυβηθεί από αυτά που ακούω για το Erasmus Plus, διότι είναι ένα project που ε, όταν έχω τα κέφια μου θεωρώ θετικό και είναι λόγος να παραμείνει η το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει νόημα και είναι και θετικά. Αλλά εάν το στρεβλώσουμε αντί ε, να είναι ο βασικός λόγος να παραμείνουμε, για μένα θα είναι ο βασικός λόγος να φύγουμε. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η παραδοχή ότι ένα είδος εθνικισμού είναι κακό και ένα άλλο είναι καλό. Δηλαδή είναι κακό να είσαι εθνικιστής με την έννοια ότι πιστεύεις στην πατρίδα σου την ίδια, αλλά είναι καλό να είσαι ευρωεθνικιστής, να πιστεύεις ότι ε, ε, ζεις σε μια χώρα εικονική που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο ένας εθνικισμός είναι καλός και ο άλλος κακός και ο υπόλοιπος κόσμος τι γίνεται. Μήπως να είμαστε λίγο πιο εξωστρεφείς. Ε, εκπαιδευτική πολιτική είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Καλέ οι βέλτιστες πρακτικές, αλλά όχι τέτοιε αποστολέ. Σε κανένα κανονισμό να μην μπαίνουν αυτά, σε καμία νομοθεσία. Και είναι κάτι που το Ηνωμένο Βασίλειο σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει έτσι Και αλλιώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις σκέψεις σας, συνάδελφε. Και τώρα ο κύριος Μαραγκάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι να πω τώρα εγώ. Ε, ε, θέλω να πω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει ο συνάδελφος Δράγκητς με την έκθεσή του ακριβώς για να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του με την οποία συμφωνώ. Τι έγινε, έχουμε ένα πρόβλημα με τη διερμηνία, κάποιο μικρόφωνο στα αγγλικά. Δεν υπάρχει διερμηνία από Ισπανικά. Βεβαίως. Εντάξει. Okay. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι συμφωνώ με τον εισηγητή και καλό είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την έκθεση και να την πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις τελικέ συνέπειες και όλα αυτά τα θετικά που μας παρουσίασε ο εισηγητής με τόσο εύγλωτο τρόπο. Συμφωνούμε όλοι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ευρώπης είναι το Εράσμος. Γιατί δεν είναι σύνταγμα, δεν είναι νόμος, δεν χρειάστηκε να εγκριθεί από εθνικά κοινοβούλια, δεν χρειάστηκε καν να ε, επιβαρυνθεί ιδιαίτερα οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα μετριοπαθές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά με τεράστια πολλαπλασιαστική αξία. Και αυτό είναι ένα πρώτο δίδαγμα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτοί οι νέοι που είναι ήδη Ευρωπαίοι, τα παιδιά και τα εγγόνια των φίλων μου και αύριο τα δικά μου τα εγγόνια, τι μας λένε. Αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες, το βλέπουμε αυτό, χωρίς να χρειάζεται τίποτα, ε, ούτε νόμοι, ούτε αποφάσεις του κοινοβουλίου υπερβολικές, ούτε τίποτα. Από την άλλη όμως δεν μπορούν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχει η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, ευρωπαϊκή ηθαγένεια, αλλά δεν καταφέραμε να τη μεταφέρουμε στην πράξη, με τη νομική έννοια, την πολιτική, τη θεσμική κτλ. Είναι μια ιδέα. Αυτό είναι ακόμα ένα έλλειμμα. Και έχει να κάνει με τις δυσκολίες ή πώς να το χαρακτηρίσω, τα εμπόδια που δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε στο παρελθόν δεν έχουμε ακριβώς εκείνο το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θέλαμε πριν από μόλις 10 χρόνια. Και καταφύγαμε, κρυφτήκαμε σε μια συνθήκη ε, βάζοντας πιο χαμηλά τον πύχη. Καταφύγιο είναι αυτό, δεν είναι. Είναι άμυνα ευρωπαϊκή και όχι κατάκτηση. Η Ευρώπη χρειάζεται ε, να βασιστεί στην ιστορία της για να προχωρήσει αν έχω να κάνω μια πρόταση, έχει γίνει και αυτή, δεν θα πρωτοτυπήσω ούτε εγώ. Αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει να αντιμετωπίσει το θέμα, το πώς θα εξηγεί στον εαυτό της την ίδια την Ευρώπη. Και κάτι που να μπορεί να είναι ε, ένα μάθημα στα σχόλια Ευρωπαϊκή Ιστορία μεταξύ μας όλοι, θα, δεν θα διδάσκει ο καθένας, δεν θα είναι η ιστορία των νικητών επί των ιτημένων ή των μεγάλων επί των μικρών ή το κέντρο απέναντι στην περιφέρεια κτλ. Θα είναι μια κοινή ευρωπαϊκή ιστορία των ευρωπαϊκών λαών και να λέμε την αλήθεια για τις ίδιες ε, τις φρικαλαιότητες και τα όσα προκαλέσαμε και πώς δεν είμαστε ικανοί να ζούμε στην ίδια Ήπειρο παρά μόνο καταστρέφοντας ο ένας τον άλλον. Ο 20ος αιώνας ήταν ε, ένα σφαγείο Θα πρέπει να το καταλάβουν οι φοιτητέ μας και οι μαθητές και να το μεταφέρουν σε ελπίδα για το μέλλον. Τελειώνω, Πρόεδρε. Σήμερα η Ευρώπη μας στέλνει μηνύματα καθημερινά. Δύο έχουμε σήμερα. Αυτή που μας έστειλε η περίπτωση της Ελλάδας, που ζητάει περισσότερη Ευρώπη, αγωνιά για να υπάρξει Ευρώπη. Πέρα και παρά τις αντιευρωπαϊκές ε, συμπεριφορές που μόλις ακούσαμε ξανά εδώ μέσα. Και επίσης έχουμε την προσφυγική κρίση που είναι άλλη κραυγή αγωνίας. Ε, ξεκάθαρη ότι χρειαζόμαστε Ευρώπη, θέλουμε να υπάρξει Ευρώπη και να φέρεται ως Ευρώπη. Όχι ως άθροισμα κρατών. Έτσι δεν είναι. Είναι, είναι, πια ορατές αυτές οι απαιτήσει σήμερα, προφανέστατες και οφείλουμε να τις μεταφέρουμε σε αξίες ε, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αυτό στοχεύει η έκθεση Ντράγκετση και θα πρέπει και εμείς να ενισχύσουμε και να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ για τις ε, σκέψεις σας. Ναι, είναι πολύ διαφορετική συζήτηση αυτή για το πώ θα δημιουργηθεί η ιστορία τη Ευρώπη, ο διάλογος για την ιστορία τη Ευρώπη. Μάλινοφ. Απλώ είναι η αρχή τη προβληματική. Γιατί ακόμα και μετά την ψήφιση και έγκριση της έκθεσης η δυσκολία θα είναι το πώς θα κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ του τι θέλουμε για την Ευρώπη και τι θέλουμε για το μέλλον της Ευρώπης και τι θέλουμε να δάξουμε στο σχολείο που είναι διαφορετικά πράγματα. Οπότε, πρώτα πρώτα να υπερμηθούμε τη κεντρική ιδέα αυτή τη έκθεση που τέθηκε ένα αμφιβόλο. Γιατί όλοι θα έχουμε πρόβλημα για να εξηγήσουμε γιατί γίνεται τούτο. Όπω διαπιστώνεται ακόμη και στην Επιτροπή μα, δεν είναι αυτονόητο. Πρώτα πρώτα υπάρχει κάποια γενική αρχή ότι μπορούμε να δούμε τι γίνεται όταν υπάρχει κάποια οργανωμένη πολιτική κοινότητα, όμως κανένα καθεστώς, καμιά κοινότητα, καμιά ένωση δεν μπορεί να το αποφύγει. Όμως είναι θεμελιώδες δικαίωμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει αυτό το ζήτημα του πώς θα διδάσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολείο. Οποιασδήποτε ένωση και φορέα είναι ε, αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή να ε, διδάσκεται ε, προκειμένου στους πολίτες και πάνω από η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι κάτι που έχει νόημα και να προσπαθεί να τους διδάξει κατά κάποιο τρόπο τον σεβασμό κάποιου είδους για να μπορούν να εκτιμήσουν αυτή την Ένωση. Αλλιώς η Ένωση και οποιαδήποτε Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στερούνται νοήματος. Οφείλουν να μην υπάρξουν εάν δεν ε, έχουν τη θέληση να κερδίσουν την έγκριση των κρατών, μελών, των πολιτών. και αυτό ακριβώς και δικαιούμεθα να προτάξουμε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχολεία. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ένωση χωρίς κάτι τέτοιο. Α τι μπορούμε να διδάξουμε στους νέους. Γιατί θα θεωρούσε ότι μια κακή προσέγγιση μπορεί να τους αποξενώσει τους νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να την κάνει κάτι το άπιαστο, κάτι το αφηρημένο όπως τώρα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό ρεύμα τώρα στην κοινή γνώμη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της ύπαρξης της Ένωσης και θεωρώ ότι το καλύτερο, και δεν το θέμα μπορούμε να έχουμε μια γενική λύση να αναδείξουν Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστορίας της συγκεκριμένης χώρας. Νομίζω ότι οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να αναπτύξει την μεθοδολογία και την προσέγγιση το ώστε να αποδειχθεί από πλευράς ιστορικής ότι είναι κάτι το καλό Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, μια κοινή προσέγγιση για όλα τα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Βεβαίως, και υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα. Ξέρουμε μεταξύ 45 και 99 ε, τι, τι σήμαινε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είχε και τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη. Άρα αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα. Επίσης, άλλο, θα πρέπει να τονιστεί όχι το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό είναι θέμα πολιτικής επιστήμης. Εντάξει, εγώ προτίθεμα να το κάνω αυτό, γιατί έχω σπουδάσει πολιτική ιστορία, πολιτική επιστήμη, οπότε μπορώ να τα διδάξω στους νέους. Αλλά η σχέση με τους νέους είναι τα δικαιώματά τους και οι ελευθερίες τους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελευθερίες και δικαιώματα. Εδώ θα βάλω μια τελεία. Αλλιώς θα πρέπει να συζητήσουμε για τα πάντα που είναι μεγάλη συζήτηση. Άρα συγκεκριμένη συσχέτιση με την ιστορία δεν νομίζω ότι κάθε χώρα έχει διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχουν δύο-τρει βασικέ γενικέ ιδέε για την Ευρώπη. Στην Δυτική Ευρώπη, δύο-τρει χώρε έχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα και από την άλλη μεριά οι πρώην κομμουνιστικέ, όπου οι περισσότερε εξ αυτών έχουν κάποια κοινού παρονομαστέ λόγω στην, στην ε, κοινή γνώμη. Αλλά και όλοι οι νέοι θέλουν να τους εξηγηθεί τι δικαιώματα και προχρώσεις έχουν, μια που, τι δικαιώματα και ελευθερίες έχουν επίσης μια που ζουν και εκείνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τους λόγους της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους πούμε και ποια είναι εναλλακτική λύση. Όχι να τους φοβήσουμε, αλλά α κάτσουν να σκεφτούν πώ θα ήταν εάν ζούσαν κάπου, σε κάποια χώρα, που δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε να δούμε πώς μπορούν να διαφυλαχθούν αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες. Και σας μιλώ από ιδία πείρα, γιατί πολύ συχνά πάω στα σχολεία στη Βουλγαρία και ξέρω πώς ε, αντιδρούν τα παιδιά. Ιστορία και ελευθερίες. Και άλλα πολλά υπάρχουν. Αλλά προσπαθώ να συμβάλλω όσο μπορώ καλύτερα στην έκθεση. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μας πιέζει ο χρόνο. οπότε οι επόμενοι ομιλητές παρακαλώ δύο λεπτά, ο κύριος και κατόπιν ο κύριος Γραμματικάκης. Word και Σεντρόβο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν μπορέσουν ε, να μεταφράσουν οι διερμηνείς αυτό που θα πω. Στη χώρα μου όμως έχουμε μια παροιμία για να δούμε αν μεταφράζεται που λέει περίπου το εξή. Ότι ε, έγινε μια μάχη για την ειρήνη και στο τέλος ε, σκοτώθηκαν όλοι. Γιατί το λέω αυτό. Ουσιαστικά η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε, αποδίδεται αυτό. Ε, ε, έχουμε την κλιματική αλλαγή, προσπαθούμε να το λύσουμε και ό,τι και να κάνουμε αυτή αυξάνεται. Στη χώρα μου τουλάχιστον όσο πολεμάμε τη διαφθορά τόσο αυτή οργιάζει. Ε, φοβάμαι δηλαδή, φοβάμαι ότι κάτι τρέχει. κάποιος το συντηρεί αυτό, το διατηρεί. Αλλιώς δεν θα υπάρχει μισθός ε, να πληρώσουμε, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να μας ε, ψηφίσουν. Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτό το μαγαζάκι να επιτίθεσαι στην Ευρώπη, ε, να έχεις αυτή την ρητορική, ποιος θα σε ψηφίσει και πώς θα σε ψηφίσουν για να βγεις ευρωβουλευτής. Αυτό είναι λοιπόν κάτι, ένα παιχνίδι που χρησιμοποιούν ορισμένοι, ένα εργαλείο που θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ε, Καλή λοιπόν η διδασκαλία ε, της Ευρώπης στο σχολείο για να έχουμε κάποιες βασικές αρχές και έννοιες που μας ενώνουν. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ε, γιατί δημιουργήθηκε η Ευρώπη. Είναι ιστορική η λόγη, πολιτισμική, γεωγραφική. Είναι ένας χώρος ενιαίος, αλλά όχι μόνο γεωγραφικά, από πάρα πολλές πλευρές. Όλοι αυτή η πολιτικοί λοιπόν σήμερα που παίρνουν ψήφους στρεφόμενοι κατά της Ευρώπης, και στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατά τα άλλα σέβομαι και τιμώ τα μάλα, γνωρίζουμε ότι τα αγγλικά είναι ένα μείγμα άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και βεβαίως και γαλλικών. Δεν υπάρχει πολιτισμός χώρα στην Ευρώπη που να μπορεί να είναι ε, αυθύπακτη και να ε, εξακολουθεί μόνη της να ε, ζει στον πλανήτη. Ούτε καμία χώρα προέκυψε έτσι ξαφνικά αναδύθηκε. Είναι με ανταλλαγές, ε, με διάφορους χώρους και γύρω από την Ευρώπη. Γι' αυτό η Ευρώπη είναι ένας ενιαίος χώρος και θα πρέπει να το γνωρίζουν τα παιδιά μας και να το μαθαίνουν στο σχολείο. Και να μαθαίνουν ότι είναι ευκαιρία να είσαι Ευρωπαίος, δεν είναι πρόβλημα. Ε, κύριος Γραμματικάκης παρακαλώ. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος ε, κυρία Πρόεδρε γιατί έχει προχωρήσει και η ώρα και γιατί όλα αυτά έχουν κουβεντιαστεί πάρα πολύ θεωρητικά στο παρελθόν. Είναι όμως απλό. Ε, η αισιοδοξία που δημιούργησαν τα παιδιά που πήραν τα βραβεία του Καρλομάγνου είναι μια οδός προς το μέλλον γιατί η Ευρώπη έχει τα τελευταία χρόνια μια τριπλή κρίση Πρώτα-πρώτα μια μακριά χρηματοοικονομική κρίση. Δεύτερο, μια κρίση που θα την η ομοιρία όλων μας στην τρομοκρατία, στις τρομοκρατικές ενέργειες, όλων μας. Και τρίτο βέβαια η τραγωδία του προσφυγικού ζητήματος που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι γνωστό. Ένα είδος απαντήσεως είναι πάντα στην ιστορία του ανθρώπου η παιδεία και ο πολιτισμός και η έκθεση του συναδέλφου Νταγκίκη, την οποία βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά πολύ δύσκολο να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα θα έλεγα ρεαλιστικό, είναι ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα σε αυτό μπορεί να δει κανένας και τη δυσκολία να γίνει ελκυστική αυτή η διδασκαλία. Η διδασκαλία συνήθως στα σχολεία αποθεί τους μαθητές. Ακριβώς όμως επειδή είναι δύσκολο και ενδιαφέρον το θέμα, για μένα προσωπικά πρέπει να προχωρήσουμε και είμαι στη διάθεση του συναδέλφου για ενδεχόμενες ιδέες και συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. κυρία Τζούλη Ward. Um, I'll be very Ευχαριστώ, θα και εγώ εξαιρετικά λακωνική, γιατί σε λίγο θα πρέπει να παρουσιάσω και τη δική μου έκθεση. Και υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, κάποιες συνέργειες μεταξύ των δύο εκθέσεων. Συνεχίζω τον ερμό του προλαλήσαντα, ε, που είπε πόσο δροσερή και υπέροχη η παρουσία των νέων το πρωί. Μα σίγουρα η Ευρώπη ανήκει στους νέους το μέλλον της Ευρώπης ανήκει στους νέους. Γι' αυτό θα πρέπει στους νέους να δώσουμε τα εφόδια και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να βρουν την ταυτότητά τους, να διερευνήσουν τις σχέσεις τους με τον άλλον, τους άλλους, Εντό τη χώρα του στι περιφέρειές του, στην πατρίδα του, στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Και επειδή εργάστηκα, απασχολήθηκα, απασχολήθηκα στην ε, μη τυπική εκπαίδευση τα τελευταία 30-40 χρόνια, ουσιαστικά είναι το έργο μια ολόκληρη ζωή για μένα το θέμα τη παιδείας. Και αυτό που χρειάζονται οι νέοι είναι βέλτιστες πρακτικέ, να μπορέσουν να διαλέξουν, να τι διαμορφώσουν στα μέτρα του, να τι αλλάξουν, να επιδράσουν σε αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με θλίβει το γεγονός όταν κάποιοι δεξιοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, νιώθουν ε, άσχημα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι Βρετανίδα, είμαι Ευρωπαία, είμαι πολίτης του κόσμου, είμαι από τη Βορειοδυτική Αγγλία, είμαι γυναίκα, έχω πάρα πολλές ταυτότητες. Και ακριβώς αυτή η η ύπαρξη των πολλών ταυτοτήτων δεν με περιορίζει, με εμπλουτίζει και μου δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό θέλω και αυτό προσπίζω για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το λέω και στην πατρίδα μου. Γιατί με λυπεί βαθύτατα το γεγονός που η κυβέρνηση δεν θα δώσει στους, κα... στους ανηλίκους κάτω των 18 το δικαίωμα ψήφου στο επικείμενο δημοψήφισμα. Γιατί παίζουμε με το μέλλον των παιδιών μας, των παιδιών των εγγόνων μας, και των φίλων των, των παιδιών των φίλων μας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή, να δώσω το λόγο στην κυρία Σόντροφ ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να διδαχθούν τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι το βασικό γιατί θα πρέπει οι μαθητές να μάθουν για τα θεσμικά όργανα, για τον τρόπο λειτουργίας τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να το παραβλέψουμε αυτό το θέμα είναι το πώς θα γίνει και αυτό πρέπει να γίνει σαν προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών κατονμερών, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς θα γίνει η δασκαλία. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο να πούμε εμείς από το Κοινοβούλιο. Το πώς θα γίνει η δασκαλία των παιδιών στο σχολείο. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι τον συντονισμό. Αυτό είναι το μήνυμα μας εμείς, αυτό προσδοκούμε από τα κράτη-μέλη. Όλοι όσοι έχουμε ζήσει στον κομμουνισμό και στις τέρες ελευθερίας έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία για οδήποτε ε, είδους ε, ιδεολογική επιρροή. Ξέρετε, στη χώρα μας απαγορεύεται να ε, γίνονται πολιτικές προκλογικές εκστρατείες Οπότε θα πρέπει να διδαχθεί η ιδεολογία, οπωσδήποτε. Και γι' αυτό σας λέω ότι αντιλαμβάνομαι το ότι πρέπει τα σχολεία να διδάξουν τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως και οι μαθητές αλλά και οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν ε, το περιθώριο να λάβουν τις αποφάσεις να διαμορφώσουν τη γνώμη τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ έχω πιστεί ότι όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, Όσο περισσότερα ξέρει κανείς, τόσο καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όμως θα πρέπει να πρόκειται περί ελεύθερης διαμόρφωσης της βούλησης της απόφασης. Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινόφ γιατί πάρα πολύ καλά μας τα είπε για το τι θα πει επιρροή. Γιατί γίνεται όταν κανείς συνεχίζει την ε, πορεία της ε, εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο. Και όπως είπε ο κύριος Μαρίνο, θεωρώ ότι όσο περισσότερο πληροφορίε, όσο περισσότερη ενημέρωση, τόσο καλύτερα. Όσα περισσότερα μαθαίνουν με χθε τόσο καλύτερε σχέσει έχουν Ευχαριστώ, συνάδελφε. Λέει πρόεδρο και τώρα να δώσουν το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν θέλουν βέβαια να μιλήσουν. Η εκπρόσωπο είναι η Σοφή Μπερνάρ. Έχετε το λόγο. Και βεβαίω και περιμένουμε να μα βοηθήσετε για να έχετε μια θετική στάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Τραγκίτση για την έκθεσή του και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση στο σεμινάριο που μας επέτρεψε ήδη να ανταλλάξουμε απόψεις. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να διδάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχολεία, αλλά κάτι τέτοιο είναι περίπλοκο και πολυδιάστατο. Γιατί δεν είναι μόνο θεσμικό, θεσμικό μόρφωμα η Ευρώπη και έχει και μια ιστορική διάσταση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, πώς θα κάνουμε τον πολίτη να νιώσει ότι ανήκει σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο. Επίσης, ε, να προωθήσουμε τις θεμελιώτες μας αξίες και αρχές. Διαπιστώσαμε από τη σημερινή συζήτηση ότι είναι περίπλοκο ακριβώς αυτό το ε, φαινόμενο και πολύ διαφορετικά το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Φυσικά θα πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους για την Ευρώπη για να τους βοηθήσουμε να διαμορφώσουν γνώμη όπως αναφέρθηκε, επίσης να έχουν τα εφόδια για να ε, δράσουν μέσα στην κοινωνία, να αναλάβουν το ρόλο τους έχοντας πλήρη γνώση της κατάστασης, να βοηθήσουμε να επιμορφώσουμε τους ε, καθηγητές για να βοηθήσουν ε, τους νέους και να τους συμπαρασταθούν σε αυτό το δρόμο. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Erasmus πλάσο η εισηγητής και σε άλλες πρωτοβουλίες, προγράμματα και πλατφόρμες ε, το, το Gateway για την ε, η διαδικτυακή πύλη για την ε, σχολική εκπαίδευση, η αδερφοποίηση και ούτω καθεξής. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες που εμπλέκουν και τους δασκάλους και καθηγητές και τους δίνει ιδέες για το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες και τους δίνει και τα εφόδια να ολοκληρώσουν τη δική τους κατάρτιση και να βοηθήσουν καλύτερα τους μαθητές τους. Πολλά εργαλεία υπάρχουν στη διάθεση των σχολείων. Θα τα αναπτύξουμε περαιτέρω για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε καλύτερα την Ευρώπη και να τη διδάξουμε λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις διαστάσεις. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής τώρα, ο κύριος Δραγκίτσι, για να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν και κυρίως αυτούς που υποστηρίζουν την έκθεση, αλλά και αυτούς που την επικρίνουν, γιατί ο καθένας ε, έχει δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του. Ευχαριστώ τον κύριο Γραμματικάκη και τον κύριο Διάπολ που αναφέρθηκαν στους νέους, ε, στους νέους που συναντήσαμε πριν από λίγο που, και που είναι ζωντανή απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όταν επισκέφθηκα το ε, όταν έφυγα από την Ρουμανία το 1989, η πρώτη ε, ε, χώρα που επισκέφτηκα ήταν η Ελλάδα. Και μερικέ φορέ μιλάω και λίγο ελληνικά με τον κύριο Γραμματικάκη. Και η πρώτη σκέψη επί Σοκράτη και, και Αριστοτέλη ήταν οι στοχαστές. Οι στοχαστές είναι αυτοί που σκέφτονται και δεν αναλαμβάνουν δράση. Ενώ οι σκεπτικιστέ, αυτό, αυτή είναι η ουσία των σκεπτικιστών ουσιαστικά. Αυτοί που απλώ στοχάζονται, κάθονται, σκέφτονται και δεν αναλαμβάνουν δράση δεν θέλω να το πάρει κανείς προσωπικά, ονόνοητο το, εν πάση περιπτώσει. Δεύτερον, κάποιος που δεν έχει μορφωθεί και δεν είναι ενημερωμένος, δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του και δεν ξέρει τι να κάνει. Εγώ ανήκω σε μία μειονότητα, του Ρωμά, και ξέρετε τι, ε, πώς δυναπαθεί η κυβέρνηση του Ρωμά, ακριβώ επειδή δεν ενημερώνεται και δεν γνωρίζει τα δικαιώματα και σκεφτείτε 500 εκατομμύρια άνθρωποι να δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του. Ένα άνθρωπο που δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του ε, γίνεται έρμεο χειραγώγηση. Είναι πολύ πιο εύκολο να το χειραγωγήσει κάποιο. Και ο Ζαν Μονέ είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν από 50 χρόνια. Είπε ότι μεταξύ των διαφορών και των, ε, και των γεωγραφικών συνόρων υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Αυτό ας μην το ξεχνούμε. Το ευρωπαϊκό όνειρο που είχαν για μας ε, ο Σούμαν και ο Μονέ. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα είναι ε, ότι ίσως η δύναμη του σκεπτικισμού και η έξαρση του σκεπτικισμού οφείλεται, ίσως λέω, δική μου πρόταση είναι ίσως, είναι γιατί μονοπολούν κάπως τη συζήτηση, ακούμε τη δική τους μόνο μουσική, δεν ακούγονται οι υπόλοιπε ε, φωνές. Και αν δεν πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα, δεν να διχαστούμε και να διαρεθούμε. Και αν κάποιος ε, είναι απολυτικός, ε, ε, ίσως θα πρέπει να μένει στο δικό του κράτος που είναι απομονωμένο ή να είναι άπατρης. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια έννοια σε εμά ότι πρώτα πρώτα είσαι πολύ καλό ηγητή πρώτα για το προσέξατε πρώτα το θέμα και δεύτερον το ότι ακριβώ επειδή προέρχεστε από τέτοια σημαντική μειονότητα του ε, Ρωμά, σημαντική για την Ευρώπη, έχετε αυτή την αποφασιστικότητα ε, σε σχέση με το πώ θα γίνει μάθημα για τα σχολεία Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε είμαι ε, σίγουρη ότι τελικά θα βρεθεί ο τρόπο να το πετύχουμε αυτό γιατί θα ράβει υπόψη μου τα περισσότερα αυτά που είπατε και για εσείς αυτά που είπατε κύριε Μαλίνοφ. Ακριβώς γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες, την ελευθερία, τα δικαιώματα, τη δημοκρατία. Θα πρέπει έτσι με την εκπαίδευση να έχουμε τον ενεργό πολίτη και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι νέοι είναι δύο ηθαγενειών, είναι και Ευρωπαίοι και ανοίγουν και στο κράτος τους. Οπότε γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο αναλφαβητισμός. Και είναι πάρα πολύ κακό το να μην συμμετέχει κανείς σε τέτοια μαθήματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Και όπως είπαν τόσοι συνάδελφοι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, κατάλληλη οργάνωση του εκδευτικού συστήματος στα κράτη-μέλη. Καλύτερες πρακτικές, ένα πλαίσιο, προτάσεις μπορούμε εμείς να τα προσφέρουμε. Γιατί η μεθοδολογία της ε, εκπαίδευσης μπορεί να είναι κοινή, τι θα κάνουν δηλαδή οι δάσκαλοι, ε, οπότε αυτό είναι δική μας υποχρέωση να το υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισήγηση. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πολύ σημαντικό. Ε, πολλά πράγματα έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Είναι έκθεση της Julie Ward για τον διαπολιτισμικό διάλογο, πολιτισμική πολυμορφία στην πρόθεση θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, όπως γνωρίζετε, ήδη για το ίδιο θέμα το Σεπτέμβριο κάναμε την ε, ακρόαση 7-12 θα ψηφίσουμε και 20 10 την Παρασκευή λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες. Τζούλι Βόρντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη Γραμματεία φυσικά και τους συναδέλφους ε, μέλη της Επιτροπής που με βοήθησαν πάρα πολύ στην έκθεσή μου. Θέλω να θυμίσω ότι η έκθεση αυτή έχει να κάνει με το ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου ε, στην προώθηση τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας κάνω μια μικρή σύνοψη η έκθεση είναι μια απόπειρα να βασιστούμε στην κοινή συμφωνία των Υπουργών Παιδείας μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Συνδυάζει τις απόψεις και τις ε, προσπάθειες που χρειάζονται για να ε, προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση ή περιθωριοποίηση και να δοθεί ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών σε όλους. Η έκθεση εντοπίζει ευκαιρίες, ιδιαίτερα μαζί με προκλήσεις βέβαια και κάνει συγκεκριμένες συστάσεις για δράση σε ε, κάθε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνει τη χρήση πολιτισμού και εξωτερικών δράσεων ε, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ανάπτυξη. Αναγνωρίζει το σημαντικό και μοναδικό ρόλο που διαδραματίζει η ε, πεδίο πολιτισμός, η ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία του πολίτη για να ε, ε, σφυλατηθούν οι κοινότητες του μέλλοντος που να είναι ισχυρές, στεναρές, θαραλές και ε, με συμμετοχή. Δύο είναι οι βασικές αρχές. Πρώτον, η σημασία να υπάρχει μια θετική αφήγηση, δηλαδή να αναγνωρίζονται οι προκλήσεις και οι δυσκολίες μεν που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά πολύ σημαντικότερο είναι να τονίζονται και οι ευκαιρίες και να παρουσιάζεται ο διαπολιτισμικός διάλογος και η παιδεία ως εργαλεία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ανέκυψε από τις συζητήσεις που είχα πραγματικά σε πάρα πολλές κοινότητες που θεωρούν ότι απειλούνται, φοβούνται. Υπάρχει ένα κυρίαρχο αφήγημα που τους αποκλείει, τους περιθωποιεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το διαλύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, να προσπαθήσουμε να είμαστε θετικοί. Ακόμα και αν προέκυψε αυτό από μια τραγωδία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Δεύτερη αρχή επίσης πολύ βασική είναι να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτό το θέμα που είναι ευρύτατο. Να μην διαχωρίζουμε την παιδεία, ε, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κτλ. Αλλά να δημιουργούμε γέφυρες και συνέργειες μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων. Η μέθοδος εργασίας ε, που με οδήγησε μέχρι εδώ ποια ήταν. Προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερες ιδέες και συνάντησα την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ, ανθρώπους που εργάζονται επί τόπου, φορείς διαφόρους. Αλλά το έκανα έτσι κι αλλιώς όλη μου τη ζωή. Δεν το εκατέλειψα όταν εξελέγει να υπερβολευτής. Αυτή τη δουλειά κάνω, ναι, καθεν. Προσπαθώ να είμαι πάντα σε μόνιμη και διαρκή τακτική επαφή με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα καθημερινά. Έχω συνεργαστεί με μέλη ΜΚΟ και τη κοινωνία των πολιτών εδώ, Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Και έχω ένα μόνιμο διάβλο επικοινωνίας με τους ανθρώπους αυτούς και με τις πιο ποικίλε ε, οργανώσεις και στο κράτος μέλος από το οποίο προέρχομαι η έκθεση μου γι' αυτό βγήκε πολύ πλούσια, βασίζεται σε στοιχεία, είναι απόρρια συζητήσεων με κανονικούς ανθρώπους ε, καθημερινούς που ξέρουν και τα προβλήματα και προτείνουν και λύσεις. Επίσης ε, συναντήθηκα με εκπροσώπους της Κομισιόν, της ε, Προεδρίας Λουξεμβούργου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαι πολύ περήφανη που έχω τη Λουξεμβουριανή Προεδρία στο πλευρό μου, έκαναν ολόκληρη διάσκεψη για αυτό το θέμα. Το καλοκαίρι ήρθαν θελοντές μαζί μου που πήγαν σε αυτή τη διάσκεψη και έτσι ε, μπορούμε να μοιραζόμαστε την εξουσία, τη λήψη των αποφάσεων με περισσότερο συμμετοχικό τρόπο. Θέλω να συμπεριλάβω όσο γίνεται τις ιδέες όλων των σκιωδών. Ήδη είχαμε μια πρώτη συνεδρίαση στην αρχή για μια γενική ανταλλαγή απόψεων και ακολουθεί δεύτερη αμέσως μετά τούτη εδώ τη συνεδρίαση, αν δεν απατώμε. Πρέπει να πάω να τσακάρω λίγο το πρόγραμμά μου ε, και σε άλλη επιτροπή έχω δουλειά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ συμμετοχική αυτή η δουλειά, πάρα πολύ παραγωγική η μέθοδος συνεργασίας μας. Κάτι που θέλω να προσθέσω για τις τροπολογίες. Βεβαίως ξέρω ότι έχουμε περιορισμό στους χαρακτήρες, στην έκταση, στο χρόνο και στο χώρο για τις εκθέσεις μας και θα πρέπει να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σύντομη και να καλύψω τα σημαντικότερα στοιχεία. Υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε πολλά σημεία, ε, αφοροποίηση στα σχολεία, πολυμορφία, συνεργασίες ε, και ε, τυπικές και άτυπες, τα θέματα του φίλου, η κληρονομιά, η ιστορία, να μην διαιρούμε, να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά. Και έχουμε και συνεισφορές μεταναστών για το πώς αντιμετωπίζουμε και προσεγγίζουμε την κληρονομιά μας την ιστορική, υπερθωριοποίηση, όχι μόνο για τις μειονότητες, να δούμε και ε, ποια είναι τα στερεότυπα, τι είναι πλειοψηφία, τι είναι μειονότητα, τι είναι πλειονότητα. Γιατί ο καθένα το βλέπει από τη σκοπιά του. Συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, ΟΗΕ, UNESCO κλπ. Και ιδιαίτερη αναφορά κάνω σε ανθρώπους με αναπηρίες, καταπολέμηση του bullying και στον κυβερνοχώρο και να εκμεταλλευτούμε απολύτως υφιστάμενα προγράμματα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να εφευρίσκουμε τον τροχό, υπάρχει η ρόδα. περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους. Προσβλέπω σε μια αγώνιμη συνεργασία και ελπίζω να βγει μια πολύ καλή έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βοηθήσει και τους Υπουργούς Παιδείας στα κράτη-μέλη για να ε, κάνουν καλύτερες πολιτικές και καλύτερα προγράμματα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω γιατί ψηφίζουμε στην Περιφερειακή Επιτροπή. Θα ακούσω όσο μπορώ, αλλά κάποια στιγμή θα φύγω τρέχοντας. Ευχαριστούμε, Ζουλή. Είμαστε σίγουροι ότι είναι εξαιρετική η έκθεση. Έχουμε λίγο χρόνο γιατί πρέπει 11.30 να έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε θα δώσω τώρα τον λόγο πρώτα πρώτα για τρία λεπτά στου σκιώδει ηγητέ και στου μη σκιώδει ηγητέ για ένα λεπτό. Ο κύριος Ολβένη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ward για την ευκαιρία που μας δίνει να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Η έκθεση βρήθη καλών προθέσεων και θα συνεχίσω τώρα στα ουγγρικά που είναι και η μητρική μου γλώσσα. Χαίρομαι που ξεκινήσαμε αυτό το έργο και μάλιστα από κοινού. Είχαμε μια πρώτη άτυπη συνεδρίαση λίγο πριν τις θερινές διακοπές. Ελπίζω να συνεχίσουμε τις ε, επαφές μεταξύ συγκήτρες και σκιωδών εισηγητών σε πιο επίσημο πλαίσιο. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε η εισηγήτρια, ότι το άρθρο 17 της Συνθήκης Λισαβόνας είναι η νομική βάση αυτής της ανακοίνωσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Έτσι έχουμε μια διαφορετική προοπτική πια για τις νομικές συνέπειες. Επίσης, όταν μιλούμε για την πρόληψη, πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό επίσης είναι να διαλέξουμε τα σωστά εργαλεία και τους σωστούς εταίρους σε αυτή την προσπάθεια πρόληψης. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη των ε, εταίρων μας, ότι το κράτος, οι κρατικές δομές από μόνες τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Χρειαζόμαστε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Και δεν αναφέρεται παρκώς και ο ρόλος της οικογένειας στην προσπάθεια αυτή. Κανένα κράτος, καμία κρατική δομή δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της οικογένειας. Μόνο ο φασισμός και ο κομμουνισμός, τέτοια καθεστώτα προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την οικογένεια. Και χαίρομαι που υπάρχει μία στο κείμενο, έχουμε και σχετική νομική βάση άλλωστε. Άλλο θέμα αφορά τους μετανάστες. Πέραν των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τις εκκλησίες, το ρόλο των εκκλησιών. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει πολύ διαφορετικές ε, νομοθετικές διατάξεις για το ρόλο των εκκλησιών και τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Θα, μπορούμε όμως να βρούμε μια, θα μπορούσαμε να βρούμε μια διατύπωση που δεν θα τονίζει τις διαφορές μας, αλλά τα κοινά μας σημεία και τις ε, κοινέ μας αξίες. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους μετανάστες. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Δεν είναι μια νέα μορφή ε, φιλοκληρισμού ή ιδεών εκκλησιαστικών. Απλώς θα πρέπει να αντιληφθούμε διαφορετικά τις διαφορές και να ανοίξουμε τις κοινωνίες μας. Λυπούμε που έχω μόνο ένα τρίλεπτο, θα καταθέσω πάντως τροπολογίες όπως είπα και στην αρχή. Βεβαίως, ο κύριος Μάουρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πολύ λακωνικός, μια και ο χρόνος μας πιέζει. Η έκθεση της κυρίας Ward είναι φιλόδοξη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που τα συζητήσαμε στην Επιτροπή και στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και μάλιστα είναι και πολύ συνοπτική και μεστή. Αξιέπαινο αυτό. Επίσης, ε, τόνισε την ανάγκη της εξωτερικής πολιτισμικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη μιας νέας πολιτισμικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Μάλιστα πρόσφατα η, η δική μου επιτροπή οθέτησε μια σχετική ε, γνωμοδότηση. Έχω μια μικρή επίκριση, με επικοδομητικό μας πνεύμα την υποβάλλω. Καλό θα ήταν να περάσουμε από το επίπεδο των ιδεών στο επίπεδο των συγκεκριμένων απαιτήσεων για παράδειγμα, να ζητήσουμε να οριστεί ένας Ευρωπαίος εκπρόσωπος ε, που θα ασχολείται με το συντονισμό και την πρόθεση των πολιτισμικών προγραμμάτων. Επίσης, ε, να προωθούμε την κοινωνική ένταξη και τον διαπολιτισμικό και δια... Ε, διάλογο. Να ζητήσουμε προώθηση των θεωρήσεων για πολιτιστικούς λόγους, ε, για εκπαιδευτικούς λόγους, υποτροφίες για δημιουργούς, ε, να λάβουμε υπόψη την ε, σύμβαση της UNESCO του 2005 και να περιλάβουμε και ένα νέο κεφάλαιο για τους μηχανισμούς προστασίας της διαφορετικότητας, της πολυμορφίας και ιδιαίτερα πληθυσμιακών ομάδων σε περίπτωση ανθρωπιστικής κρίσης για να ταχθούμε υπέρ μιας ευρωπαϊκής και οικουμενικής ηθαγένειας προωθώντα το πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή Ευρώπη και Πολίτε, για τον οποίο έχω και γνωμοδότηση, Προωθώντα την αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. Ελπίζω να συμβάλλω και εγώ με τις τροπολογίες μου στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ κύριος Μαραγκάλ και μετά κύριε Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη πρόκειται να συντάξουμε κάποιες τροπολογίες. Και όλες όμως θα είναι υπέρ ούτως Δεν θα είναι για να πούμε κάτι αντίθετο ή να αλλάξουμε κάτι. Θα είναι για να προσθέσουμε κάτι, μια διευκρίνηση, μια προσθήκη. Να διευκρινίσουμε επομένως κάποια από αυτά τα σημεία. Mm, ναι, ναι, τα είπαμε όλα για να δούμε το πώς θα τα υπενθυμίσουμε και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το οποίο λέει ο χάρτης των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων που συνεχίζει να ισχύει. Αλλά όμως θα πρέπει να το αναδεικνύουμε. Αυτό για την κοινή ευθύνη και υπευθυνότητα όλων των δημοκρατιών και δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και των ε, ΜΜΕ, των πολιτικών κομμάτων κλπ. Και αυτό θα πρέπει να τονίσουμε το ρόλο τους. και ότι η πολυμορφία των κοινωνιών μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα ΜΜΕ. Επίσης για το πώς καθηγητές και δάσκαλοι θα μπορέσουν να γίνουν φορείς της αναγνώρισης της ε, πολυμορφίας και πολυπολιτισμικότητας. Επίσης, για το ότι θα πρέπει κάπως όλα αυτά να είναι δεσμευτικά. Η απαγόρευση της δεσμενούς διάκρισης και έτσι να πρετανεύει η πολυπολιτισμικότητα. κυβερνούσε όλα αυτά να είναι εντεταγμένα στο εθνικό δίκαιο για να έχουν άμεση εφαρμογή. Επίσης, σε συνέχεια των όσων είπαμε και προηγουμένως, θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς θα χρησιμοποιηθεί το έρασμος ή κάτι σαν το έρασμος για καθηγητές και δάσκαλους για ε, δημοτικά και για γυμνάσια να υπάρχει μια τέτοια ανταλλαγή δασκάλων και καθηγητών το οποίο θα είναι προστιθέμενη αξία η πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, διαβάζοντας την έκθεση αυτή, λέω ότι ακόμα και αν το όνειρο έγινε φιάλτης, ορισμένοι από εσά δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα με τον ίδιο αγγελικό τρόπο και δογματικό τα βλέπετε, με καλές προθέσεις και με μανία αρνείστε την πραγματικότητα. Μιλάτε για την πολιτισμικότητα με ιδεολογία. Όταν το 10 και το 11 η Μέρκελ και η Κάμερον όταν προσπάθησαν να εφαρμόσουν στις χώρες τους ε, ομολόγησαν και αναγνώρισαν ε, την αποτυχία αυτής της ωραίας θεωρίας. Διαβάζοντας την έκθεση διαπιστώνουμε ότι αυτό που σας διέπει είναι παγκοσμιοποίηση ως ιδεολογία παρά η πραγματικότητα. Τρομοκρατικές επιθέσεις, πολλαπλές έγιναν στα κράτη-μέλη. Βλέπετε τη ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό Ποιος στέει, οι κακοί λαοί της Ευρώπης που αποκλείουν τις μειονότητες από τη λήψη των αποφάσεων και από την κοινωνία και χειρότερο ορισμένοι ε, ε, επικαλούνται και την ιστορία τους, λέει, για να διχάσουν. Μα η ευρωπαϊκή λαοί, κυρία εισηγήτρια, είναι οι αποκλεισμένοι και οι απόκληροι. Σε εκείνους ζητάτε να υποστούν τα κύματα των μεταναστών και να πανηθούν την ιστορία τους. Είναι ένας δούριος ύπος αυτών ε, των ε, ευρωμακαρίων που προσπαθούν να επεκτείνουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης εις βάρος των κρατών μελών. Οι πατριώτες βουλευτές που προσπαθούν να φέρουν ε, λίγο ρεαλισμό να διηθήσουν σε αυτό το κείμενο αποτυχάνουν και θα το καταψηφίσουν. Πλουραλισμός στον πολιτισμό. Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε οπότε και εγώ τώρα να δώσω το λόγο για ένα λεπτό στους υπολείπους που δεν είναι σκιώδες ehm, Και συμπαράτε με γιατί τέλειωσε ο χρόνος, οπότε τι να κάνουμε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, αλλιώς θα, θα ε, παράγουμε τελείως τα χρονικά όρια. Νέκοφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καμία χώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει μόνη της αυτήν την ε, κρίση. Παγκόσμια κρίση, παγκόσμια και λύση. Και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το μεταναστευτικό ε, και έχουμε αυτό, αυτές τις ε, προτάσεις του Γκάμπριελ και Μίλιμπαν. Πιστεύω ότι κάθε επιμέρους πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε κάποιες αξίες, ότι για τους νέους η κινητικότητα, απασχόληση, εξωτερική πολιτική, και για τη ισότητα ανδρών γυναικών, όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Χρειαζόμαστε κάποιες διαδικασίες ολοκλήρωσης και στην παιδεία, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θα πρέπει όλα αυτά να αναφερθούν στην έκθεση. Και εμείς, σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τον διαπολιτικό διάλογο και την διαπολιτιστική διπλωματία, ούτω ώστε να αναπτυχθεί η εξωτερική μας πολιτική και οι άλλες πολιτικές της Ένωσης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάποιους ε, φόβους, φόβους ε, θρησκευτική, εθνική ε, επικράτησης, άρα θα πρέπει να γίνει αυτό με εκπαίδευση και θα πρέπει όσο γίνει πιο νωρίς στο σχολείο να αυτές οι νέες αξίες να ανακρίνονται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο. Η σημερινή συζήτηση ε, και για την έκθεση του αλλά και για την έκθεση Γκόρτ ε, δείχνει σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο θεμάτων και της ε, σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ακούσαμε τα επιχειρήματα από τους συναδέλφους και ακούσαμε ότι έχουμε και νομικά μέσα στη διάθεσή μας που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και νομική βάση ε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ακούσουμε για να κατανοήσουμε. Γι' αυτό έτσι θα έχει, το, το... έτσι νόημα ο διάλογος. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα στρατευμένος και προσυλλομένος στο θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι μόνο με το διάλογο ε, και το διαπολιτισμικό διάλογο θα προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή, αλλά θα πρέπει από κοινού να βρούμε θετικές και καλύτερες λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι, ε, μιλώ εξ ονόματος του καθηγητού Βρέσκη που είναι ο Σκιώδης. Ρασναντεύσκη. Είπαμε ότι δεν πρέπει να επανεφεύγουμε τον τροχό, είπε κάποιο. Κοιτάξτε, υπάρχει βικουρικότητα εδώ που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι άλλο είναι να καταλαβαίνει κάτι και άλλο να λες ότι όλα είναι όμορφα, ηθικά, εγκεκλικά πλασμένα και η κάθε ομάδα είναι τέλεια. Αυτή η συζήτηση συνδέεται και με προηγούμενες. Ελπίζω να μην υποθέσουμε ότι όσοι διαφωνούν δεν κατανοούν την ιστορία κατά κάποιο τρόπο ε, ή δεν τρώνε διαφορετικά φαγητά. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι αλαζονικά πράγματα και δεν χρειάζεται να τα σχολιάσω. Ακούστε παρακαλώ τις δημοκρατικές φωνές με τις επιφυλάξεις και το σκεπτικισμό γιατί αν τις αγνοήσετε οι εναλλακτικές λύσεις μπορεί να είναι πολύ χειρότερες. Ευχαριστώ. Eh, νομίζω ότι συμφωνούμε. Και τώρα γραμματικά έχει την τρούπελ. Σύντομα. Και εγώ όπως πάντα ε, νομίζω ότι το θέμα που προσπαθεί να θίξει η έκθεση είναι απέραντο. Περίπου όπως το ίδιο το σύμπαν και πρέπει να αποφύγουμε λίγο τις μαύρες τρύπες από αυτά που διάβασα νομίζω ότι η κυρία Γουόρτ κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αναδεικνύει πραγματικά τα σημαντικά θέματα που εγώ θα ήθελα να γίνουν λίγο περισσότερο πρακτικές οι προτάσεις και επίσης θα ήθελα στην έκθεση να αναδειχθεί με ευγενικό τρόπο ότι η απόσταση, το λέω συχνά κυρία Πρόεδρε, των λόγων από τις πράξεις στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και ενώ όλοι ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στην πολυμορφία, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, σε αυτά τα θεμελιώδη αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πράξη, όπως για παράδειγμα το τελευταίο πακέτο Juncker που αγνοεί περίπου συνολικά αυτές τις αξίες, είναι διαφορετική και θα ήθελα να αναδειχθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κάτι να πω στον συνάδελφο από την Γαλλία. Γιατί νομίζω. Τι συνάδελφο από την Γαλλία μου. Γιατί πο, ποτέ δεν ήταν ει βάρο εθνική ε, ε, ταυτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνυπάρχουν. Αυτό ακριβώ είναι ο πύρινο του θέματο. Δεν σα αποστερούμε αυτή την ταυτότητα. Πρόκειται ακριβώ για εμπλουτισμό, Πρόκειται για κάποιους χειραφέτηση και επίσης θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή την έκθεση. Η πολυμορφία και ο διάλογος ο διαπολιτισμικός. Γιατί η εξωτερική πολιτική θέλει να προλάβει την βία, η ιστορική πολιτική αφορά την κατοχήρωση κάποιων θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και του χρόνου θα πρέπει να ανανεωθεί ούτως επίν το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον διαπολιστικό διάλογο και αυτό όμως πρέπει να αναδειχθεί μέσα από την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Προηγουμένω δεν σα δόθηκε ευκαιρία να μιλήσετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είμαι σύντομη. Θα ήθελα απλώ να πω ότι ε, υπό τη σκοπιά της εκπαίδευσης, γιατί έχουμε και τη σκοπιά του πολιτισμού, ή θεωρούμε την έκθεση πολύ καλή και επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία και τονίζει τη σημασία τους. Είναι πολύ επίκαιρη άλλωστε η έκθεση και είναι συμβατή ε, και με τη διακήρυξη των Παρισίων των Υπουργών Παιδείας. Πολύ θετικό αυτό. Επίσης η έκθεση αναφέρεται στα διάφορα επίπεδα της παρέμβασης, το κρατικό και το ευρωπαϊκό, όπως προβλέπει και η ίδια η διακήρυξη των Παρισίων. Επίσης, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και πραγματικά η ε, έκθεση γεφυρώνει την εκπαίδευση με τον διαπολιτισμικό διάλογο. Και είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε διατομιακή προσέγγιση για τα θέματα αυτά. Δύο τώρα συγκεκριμένα σχόλια. Ίσως ε, το κείμενο θα πρέπει να είναι πιο σαφές και πιο συγκεκριμένο για το είδος των ε, προσεγγίσεων που θα χρησιμοποιήσουμε στην παιδεία για να προωθήσουμε την διαπολιτισμική κατανόηση. Επίσης, ε, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα έχουν ρόλο κλειδί στην προσπάθεια αυτή. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, τη διατύπωση για το ρόλο τους. Και επίσης στο επεξηγητικό σημείο μας στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεστε πολύ σωστά στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Ίσως θα πρέπει να αναφερθείτε και στο πλαίσιο πολιτικών που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την επαγγελματική κατάρτιση για το 2020 και την επιμόρφωση Οπότε καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε από κοινού το Erasmus Plus και το, την επιμόρφωση 2020 για να δώσουμε μια συνέχεια στην διακήρυξη των Παρισίων. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρησιμοποιητά. Ευχαριστώ όλους. Το Δικαίωμα θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και για τις τροπολογίες έχουμε προθεσμία ε, στις 23 Οκτωβρίου. Όπως είπε η Επιτροπή. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση γιατί αναδεικνύεται ο ρόλος της παιδείας και κάποιες αξίες που είναι κοινέ. Και βοηθάτε έτσι ο διαπολιτισμικός διάλογος, κάτι το οποίο δεν αφαιρεί αλλά προσθέτει. Είναι η αλληλοκατανόηση. Και όπως τα είπατε και εσείς, Έχουμε τώρα την κρίση σε πολλά μέτωπα και για τον, γεωπολιτικό ε, διάλογο και για άλλα. Όλα αυτά επομένως θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και έτσι να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να γίνει αυτή η πλαισίου στην παιδεία οπότε να ξέρουμε τι γίνεται, να βοηθήσουμε τους ε, δάσκαλους όπως τα είπε και η συγκίδρια Word. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τελειώνει η πρωινή συνεδρίαση και θα αρχίσει και κλεισμένο να η συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ συνάδελφοι, εσείς που είστε εδώ, ελάτε και το απόγευμα που αρχίζει στις 3 δημόσια ακρόαση όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης σε συνεργασία και με την Επιτροπή πολιτικών ελευθεριών. Πολύ σημαντική η ακρόαση. Ελπίζω να έρθετε. Πολύ ενδιαφέροντος είναι και προσκεκλημένοι μας. Οπότε παρακαλώ ε, γρήγορα αποχωρήστε όσοι πρέπει γιατί ήδη είμαστε πίσω από το χρονοδιάγραμμα γιατί τώρα αρχίζει και κλεισμένων συνεδρίαση των εισηγητών. Thank you because we need to begin